Excellencies. Εξοχότατη. Excellencies, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, έχω τη μεγάλη χαρά να σας καλωσορίσω στο φετινό στη φετινή συνδιάσκεψη της Exa World και Jean Monnet. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε απόλυτη ησυχία για να ξεκινήσει μουσικά η συνδιάσκεψη αυτή από την κυρία Ναταλή Νικό, μια σοπράνο με εξαιρετική φωνή και διεθνή καριέρα, η οποία θα ερμηνεύσει για μας την Οδύστη Χαρά. Η κυρία Ναταλή Νικό. Κύριε Νικό, εκ μέρου όλων των συμμετεχόντων θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά πολύ για αυτή την εξαιρετική μουσική εισαγωγή στι σημερινέ μας δραστηριότητες. Κύριε και κύριοι, Τώρα έχω το προνόμιο να σας παρουσιάσω τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, ξέρω από προηγούμενες ε, συνεδριάσεις Jean Monnet και από συμμετέχοντες πόσο έχουν εκτιμήσει την διαθεσιμότητά σας να βρείτε χρόνο να, ήρθε, να είστε παρόν και να μας ε, κοινοποιήσετε και τις ε, ε, απόψεις σας. Είναι σχεδόν μια μόνιμη τιμή κατά κάποιο τρόπο για μας και για μια ακόμη φορά σε αυτή την αίθουσα θα έχουμε και τη χαρά και το προνόμιο να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τις απόψεις σας για την συνθήκη της Λισαβόνας και την εφαρμογή της. Κύριε Πρόεδρε, σας καλώ να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, τα εισαγωγικά. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι Ανδρούλα, είναι χαρά για μένα να σας καλωσορίζω σήμερα εδώ, ειδικά τους καθηγητούς, καθηγητές Ζωμονέ που ήρθαν στις Βρυξέλλες από ολόκληρο τον κόσμο και να ξεκινήσω αυτή την ε, ε, εναρκτήρια συνεδρίαση με τον πρόεδρο της Επιτροπής, της Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Ε, ξέρετε πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή σας σε αυτό το δημόσιο φόρουμ σήμερα. Το δίκτυο Ζωμονέ είναι μια τεράστια ε, κοινότητα γνώσης ε, ε, και έχει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο πραγματογνωμοσύνης. Με παρούσα σε 62 χώρες, σε 5 υπήρους και δίνεται ορατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμια και συμβάλλεται σημαντικά στις πανεπιστημιακές σπουδές για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Παράλληλα, είστε όμως ανεξάρτητοι είστε ε, επικριτικές φωνές ε, και ακριβώς ε, γι' αυτό το λόγο οι απόψεις σας γίνονται σεβαστές και είναι το καλύτερο όπλο εναντίον οποιασδήποτε δημοκοπικής κατά κάποιο τρόπο και λαϊκίστικης φωνής. Θα ήθελα να σας καλέσω να σας καλέσω να διατηρήσετε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Πρόταγμα. Ε, βεβαίως, ε, παρόλη την ανεξαρτησία, είμαστε σε φάση ακριβώς να χρειαζόμαστε αυτές τις ανεξάρτητες πληροφορίες και συμβουλές που μπορείτε να δώσετε. Ε, ακούμε προσεκτικά... Ε, ε, τις απόψεις σας, ειδικά το γραφείο των ε, Ευρωπαϊκών, των Συμβούλων Ευρωπαϊκών Φορέων ε, με πρόσωπο τον Jean-Claude που συνεργάζεται πολύ μαζί μας και είναι εδώ σήμερα μαζί μας ε, και δίνεται πολύ μεγάλη συνεισφορά, ε, αν θέλετε βέβαια, στην διαμόρφωση πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, είναι παράδοση για μας να χρησιμοποιώ αυτή, αυτό το φόρουμ για να μιλήσω για βασικές εξελίξεις. Πέρσι μίλησα σχετικά με το πώς άλλαζε τον κόσμο η παγκόσμια οικονομική κρίση. Μίλησα για την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια πιο πολιτική Ευρώπη και κάλεσα τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν την αλληλεξάρτησή τους και να δεσμευτούν περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φέτος όντως, δημιουργούμε μια πιο πολιτική Ευρώπη και η έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα μπορεί να συμβάλλει σε αυτό και συμβάλλει σε αυτό. Ε, αυτό είναι το θέμα της φετινής συνδιάσκεψης και θα ήθελα να σας πω κάποιες από τις απόψεις μου σχετικά με το τι σημαίνει αυτό σήμερα, τουλάχιστον από την οπτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τη δική μου οπτική γωνία σχετικά με το τι συμβαίνει στους ευρωπαϊκούς φορείς. Όπως ξέρετε, η οικονομική κρίση δεν έχει περάσει. Θα πω δύο λόγια όμως για τι φιλόδοξες ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχύσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Τα κράτη-μέλη δηλαδή θα δεσμεύονται και πολιτικά σε, περισσότερο σε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά ας μιλήσουμε πρώτα για την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν χρειάζεται να σας πούμε το περιεχόμενο. Ε, εξάλλου είστε όλοι καλύτεροι γνώστες από μένα. Ε, πάντως θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Όπως ξέρετε, η Ευρώπη ήταν πάντα μια ενιαία αγορά. Η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο πείραμα πολιτικής ολοκλήρωσης στον κόσμο. Είναι μια κοινότητα νόμου και αξιών και αλληλεγγύης. Ε, οι, ισχυροί δεσμοί, ισχυροί θεσμοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορούν να εφαρμόσουν διάφορες πολιτικές που είναι όλες ευρωπαϊκού περιεχομένου. Είμαστε όλοι κληρονόμοι, αν θέλετε, αυτού του δώρου και οραματιστές πολιτικοί θέλουμε να γυρίσουμε τη σελίδα του παρελθόντος. Οπότε με ξαφνιάζει που ορισμένοι ερμήνευσαν τη συνθήκη της Λισαβόνας ως ήττα ε, για την ε, ευρωπαϊκή ενοποίηση και ως ε, νίκη του ομοσπονδιακού μοντέλου. Τίποτα όμως δεν μπορεί να είναι πιο μακριά από την αλήθεια. Θα δείτε ότι ε, ουσιαστικά έχουμε περισσότερη ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και όχι λιγότερη. Ενισχύει και εφαρμόζει, θέτει σε εφαρμογή όλ, όλους τους φορείς. Παρέχει νομιμότητα στις αποφάσεις μας. Ε, όλες οι νομοθετικές πράξεις πλέον ε, ε, εγκρίνονται με συναπόφαση με την ειδική πλειοψηφία, ειδικά στα εσωτερικά θέματα θα πούν ορισμένοι ότι η ειδική πλειοψηφία κατά κανόνα σημαίνει περισσότερο διακυβερνητικό μοντέλο και λιγότερο κοινοτικό αλλά ε, ο ανισχυμένος ρόλος του Κοινοβουλίου που εκλέγεται από τους πολίτες σημαίνει ε, περισσότερο διακυβερνητικό μοντέλο και λιγότερο κοινοτικό. Ε, οι νόμοι εγκρίνονται με αυτόν τον τρόπο, αποκτώνται νέες ε, ε, αρμοδιότητες ειδικά στα οικονομικά νομισματικά θέματα και στα εξωτερικά ζητήματα. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι η ύπατος εκπρόσωπος είναι και αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Αυτό δείχνει ε, ότι συγχωνεύονται τρεις προηγούμενοι κανόνες ώστε να αποφεύγουμε σύγχυση και πολυφωνία και τα εξωτερικά εργαλεία χρησιμοποιούνται πλέον και για την ανάπτυξη πολιτικής και την εκπλήρωση πολιτικής. Κάτι το οποίο έκανε παλιά ο ύπατος εμπρόσωπο, ένα μέλος της Κομισιόν και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Τώρα αυτά γίνονται από ένα άτομο. Η νέα υπηρεσία εξωτερικών θεμάτων που έχει την ευθύνη της ε, ε, διπλωματίας ενισχύει το ρόλο και τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Ε, να συνοψίσω ένας νέος μόνιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο συμβάλλει στην ενίσχυση της, Ευρώπη της Ευρώπης μέσω συνέχειας και ισχυρότερης ηγετικής ε, στάσης στο Συμβούλιο βλέπουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως αντίπαλο της Κομισιόν, εμείς τον βλέπουμε ως ένα ισχυρό σύμμαχο, ο οποίος μας βοηθάει να συμβάλλουμε, να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό πρόταγμα, αν υπάρχει βέβαια καλή συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων και από την εμπειρία που έχω από τα τελευταία έξι χρόνια στη θέση αυτή, το βασικό πρόβλημα που έχουμε όταν ε, μιλάμε για απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόβλημα δεν προκύπτει από, τα, από τους θεσμούς, από τα όργανα, εάν τηρούν τις αρμοδιότητες και ε, εμπνέονται από το ευρωπαϊκό πνεύμα. Όχι, τα προβλήματα προκύπτουν από στενόμυαλους και εθνικιστές πολιτικούς ε, ηγέτες σε εθνικό επίπεδο. Πώς αυτά τώρα θα ισχύσουν είναι ένα μεγάλο βήμα και σαφώς υπάρχει μεγάλη πρόκληση. Θέλουμε περισσότερη ευρωπαϊκή προσέγγιση και πιο κοινή ευρωπαϊκή δράση και έτσι πρέπει να είναι διότι όταν ακολουθούμε μια κοινωτική προσέγγιση με βάση το σεβασμό των αρμοδιοτήτων όλων των οργάνων και έντιμη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και οργάνων μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Τώρα θα ήθελα να σας πω πώς ε, θεωρώ ότι ορισμένοι παρερμήνευσαν την, την συνθήκη της Λισαβόνας, διότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στην ε, αλλαγή αυτή. Η, ε, η, η συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει αυτή την πολιτική βούληση, διότι χωρίς αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί τίποτα. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας θα είναι πιο αποτελεσματική, πιο δημοκρατική και πιο ορατή σε παγκόσμιο επίπεδο και αντί να είναι η έμφαση στην οικονομική ε, οργάνωση, η ε, συνθήκη της Λισαβόνας φαίνεται ότι γίνεται ένα τελευταίο, αν θέλετε, λιθαράκι σε μια Ευρώπη που γίνεται όλο και πιο ενωμένη. Τα ε, κράτη-μέλη ε, θα δεσμευτούν περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα αναγνωρίσουν την αυξανόμενη αλληλεπίδραση. Τώρα, ε, η πρόταση της Κομισιόν για περισσότερη ε, για μεγαλύτερη και καλύτερη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Ε, κάτι που ανέφερα πριν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί και το ευρώ και οι ευρωπαϊκές οικονομίες χτυπήθηκαν. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ε, ανάπτυξη και χωρίς ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος από την ε, κρίση, ούτε επενδύσεις και ούτε ευημερία για, τις, για τους πολίτες. Ε, χτυπηθήκαμε από την κρίση στην Ελλάδα και γιατί είναι αλήθεια ότι είναι αλήθεια βέβαια ότι η επιδείνωση στα δημόσια οικονομικά προσπαθεί μας έχει υποχρεώσει να ε, αυξήσουμε την ενίσχυση για να χτυπήσουμε την κρίση, ε, αλλά υπάρχει και ένα θέμα διακυβέρνησης. Ναι, γίνονται κερδοσκοπικές προσπάθειες, αλλά το κερδοσκόποι ε, ουσιαστικά σερφάρουν και σε, ένα, κύμα και το κύμα αυτό είναι μεγάλα ελλείμματα και έλλειψη μεταρρυθμίσεων. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δίνουμε στους ε, κερδοσκόπους τη δυνατότητα να σερφάρουν σε αυτό το κύμα και ε, ε, υπάρχει μια παρερμηνία, δηλαδή η πραγματικότητα παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα της δράσης των κερδοσκόπων ή ως έλλειψη, ως αποτέλεσμα έλλειψης μεταρρυθμίσεων. Να το θέσω ξεκάθαρα. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό που θα πω. Πολλά κράτη-μέλη δεν έκαναν τις διακτροτικέ μεταρρυθμίσεις που χρειάζονταν και δεν τήρησαν ε, το σύμφωνο σταθερότητας και τις αρχές της ε, οικονομικής σταθερότητας που βρίσκονται εγγεγραμμένες ε, και στη συνθήκη της Λισαβόνας αλλά και σε προηγούμενες συνθήκες. Και η κρίση έδειξε ότι χρειάζονται περισσότερο μέτρα και τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί για να καλύψουν τις ανισορροπίες δεν ήταν επαρκή. Και βεβαίως πρέπει να δούμε τώρα τι θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση μη τήρησης των συνθήκων. Όπως η κρίση των τραπεζών, αυτή η κατάρρευση της εμπιστοσύνης έδειξε πόσο αλληλένδετα είναι οι οικονομίες της Ευρώπης και μια κρίση σε ένα κράτος μέλους μπορεί να επηρεάσει όλα τα άλλα κράτη και όχι μόνο στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις παγκόσμιες αγορές. Αν χρειαζόταν κάποια περισσότερα επίπεδα, ε, κάποια περισσότερη απόδειξη για το επίπεδο αλληλένδετα αλληλοσύνδεσης ε, δείχνει αυτό ε, ότι ε, το ευρώ είναι μια τρανή απόδειξη της αλληλοσύνδεσης που έχουμε μεταξύ μας. Και βεβαίως όλα αυτά ισχύουν και στην Ευρωζώνη και για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήρθε η ώρα να ενισχύσουμε το ε από το, το οικονομικό στοιχείο, δηλαδή από την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Όπως είπα, δεν μπορούμε να έχουμε νομισματική ένωση χωρίς οικονομική ένωση. Στις 7 Μαΐου του 2008, όταν παρουσιάσαμε την έκθεση των πρώτων 10 ετών του ευρώ, ε, Πολύ ρητά είπαμε ότι ήταν επιτυχία το ευρώ, αλλά για να συνεχίσει να είναι επιτυχία χρειαζόμαστε ισχυρότερη, ισχυρότερο οικονομικό συντονισμό, ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη και αντιμετώπιση κάποιων ισορροπιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Δύο χρόνια μετά, τα κράτη-μέλη κατάλαβαν, πιστεύω, ότι έτσι είχαν τα πράγματα και κατά κάποιο τρόπο ε, τι προτείνουμε να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης τηρούνται. Ε, δηλαδή, έλεγχος των ε, προϋπολογισμών των κρατών μελών θα διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα τηρούν τους κανόνες. Κάποιοι ε, έχουν αντίρρηση με αυτή την πρόταση της Κομισιόν, διότι επικαλούνται την αρχή της κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας. Ε, είναι σαν να μην αναγνωρίζουμε την απλή πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα κράτος μέλος θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική πολιτική και κατάσταση όλων των άλλων κρατών μελών. Και όπως το αναγνωρίζει και η συνθήκη της Λισαβόνας, η οικονομική πολιτική ενός κράτους μέλους δεν είναι απλώς θέμα εθνικού συμφέροντος ή ενδιαφέροντος. Είναι θέμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επομένω έχει νόημα να ενισχύσουμε Ουσιαστικά ενισχύονται οι αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβουλίων που συνδέονται με άλλα κοινοβούλια όταν προετοιμάζουν τους προϋπολογισμούς τους. Διότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα κοινοβούλια και οι δικές μας αποφάσεις έχουν αντίκτυπο σε όλη την, Ευρωπαϊκή, την Ευρωζώνη αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής. Πρέπει να δούμε όμως πώς ε, αντιδρούν κάποιοι πολιτικοί ε, εναντίον κάποιου θέματος το οποίο είναι κοινού νου, ε, κοινής λογικής. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι η απόφαση του Κοινοβουλίου της Ελλάδας, ας πούμε, θα έχει αντίκτυπο στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, στην, ε, στο Γαλλικό, στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, θα έχει αντίκτυπο σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει νόημα λοιπόν από πολιτικής και θεσμικής απόψεως να γίνει αυτή η αξιολόγηση ομοτήμων αν θέλουμε να έχουμε σταθερότητα και ευημερία στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα πρέπει να δούμε τις πολιτικές αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δημιουργήσουμε μια νέα αγορά για το μέλλον που να παράγει, να δημιουργεί ε, αηφόρες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Και πάντα εξετάσαμε την πολιτική ε, στην έκθεση και το φθινόπωρο που κάναμε τον απολογισμό του προγράμματος σταθερότητας και σύγκλησης. Αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να εξετάζουμε τις πολιτικές και τις επιπτώσεις του στην δημοσιονομική πολιτική ταυτόχρονα. Γι' αυτό το λόγο είπαμε να δημιουργήσουμε ένα ε, εξαμηνιαίο πρόγραμμα ε, όπως προέκυψε τώρα από την κρίση για να μπορούμε να παρακολουθούμε τους προϋπολογισμούς. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ανισορροπίες που οδήγησαν στην κρίση και είναι ακριβώς ε, ανάγκη να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση ώστε να εξετάσουμε όχι μόνο τις μικροοικονομικές πτυχές, τις μακροοικονομικές, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την εξωτερική διάσταση. Δεν μπορείς να έχεις μια οικονομική πολιτική για την Ευρώπη που να είναι τόσο κατακαιρματισμένη σαν να μην ζούσαμε στον ίδιο κόσμο, σαν ε, να μην έπρεπε να λάβουμε υπόψη τις διάφορες πτυχές και τις επιπτώσεις που έχει η οικονομία μας και η ανάπτυξή της. Δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουμε την εθνική κυριαρχία και θα αναλάβουμε εμείς τα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών. Θέλουμε όμως να υποφεληθούν τα κράτη-μέλη από την ανάλυση που θα κάνουμε του προπολογισμού τους και των οικονομικών επιδόσεών τους. Προφανώς, εάν δεν ληφθεί διορθωτική δράση, δεν θα, μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και τις κυρώσεις. Κανένας δεν, σε κανένα δεν αρέσουν οι κυρώσεις. Εγώ είπα να τις αποκαλέσουμε κίνητρα για συμμόρφωση. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται να δώσουμε αξιοπιστία στους κανόνες. Αν δεν δώσουμε αξιοπιστία στους κανόνες μας, πάρα πολύ πιθανό δεν θα τηρηθούν οι κανόνες μας. Γι' αυτό το λόγο τώρα προτείνουμε και κάποιες κυρώσεις. Όχι με την ιδέα να τις εφαρμόσουμε, αλλά να δώσουμε κάποια κίνητρα στα κράτη-μέλη, να εφαρμόσουν τα διορθωτικά μέτρα, ώστε να μην χρειαστεί να ε, επιβάλλουμε αυτές τις κυρώσεις. Θα ήθελα τώρα να είμαι σαφής. Δεν ε, θα πάρουμε τους οικονομικούς πόρους από τα κράτη-μέλη, ειδικά όταν βρίσκονται σε δυσκολίες. Αυτά που λέμε όμως είναι ότι θα πρέπει να δούμε πώς μετά το 2013 οι προϋπολογισμοί θα καταρτίζονται τηρώντα του κανόνε και τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανώνται τα χρήματα. Φυσικά η πρόληψη είναι καλύτερη από τη διόρθωση, αλλά ακόμη και αν οι διορθώσει δεν είναι αρκετέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τα μέσα να αναλάβει άμεση δράση, να μπορεί να παρεμβαίνει πιο νωρί σε μια κρίση, αυτή τη στιγμή θα έχουν αποτύχει και η πρόληψη και η διόρθωση. Τότε χρειάζεται περισσότερη δράση και όχι τόσο αντίδραση. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε ένα σταθερό πλαίσιο για τη διαχείριση των κρίσεων. Και όταν διαβάζετε, αν διαβάσατε τις εφημερίδες τους τελευταίους τρεις μήνες, θα, θα μπορούσαμε να σας συγχωρήσουμε για την άποψη που μπορεί να σχηματίσατε για τη συνθήκη της Λισαβόνας, ότι η ε, σταθερότητα του ευρώ είναι ο μόνος μας καημός και η μόνη μας ανησυχία. Ε, προσπαθήσαμε να αποφύγουμε την κατάρρευση της Ελλάδας και να στηρίξουμε την Ευρωζώνη. Κάναμε ένα πρόγραμμα με τις αρχές της Ελλάδας. Δώσαμε ένα δάνειο το 2010 ε, κάποια δισεκατομμύρια ευρώ ε, βοήθεια στην Ελλάδα και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, μία από τις χειρότερες κρίσεις που αντιμετώπισε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και κατά ορισμένου την χειρότερη κρίση που συνέβη ποτέ, διότι ήταν πραγματική δοκιμή και για τη συνθήκη και για τους κανόνες και για την αρχή της ε, Ευθύνη και αλληλεγγύης. Η κρίση όμως δυστυχώ αυτή δεν έχει περάσει ακόμα και εξακολουθούμε να βρούμε την καλύτερη διέξοδο. Το σαφές όμως είναι ότι αν βρούμε, το να βρούμε μάλλον τη σωστή κατεύθυνση είναι ευκολότερο με τη συνθήκη της Λισαβόνας και επανέρχομαι στο θέμα. Είναι απλό ότι με το νέο άρθρο 136, χωρίς, αυτό, δεν θα μπορούσαμε να προτείνουμε την ενίσχυση της εποπτείας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Βασιζόμαστε με το, στο άρθρο 136 και έτσι η Κομισιόν θα υποβάλει τις προτάσεις οι οποίες πληρώντας τις προϋποθέσεις της συνθήκης θα ενισχύσουν τη διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι πιο δύσκολο τα, τα πράγματα, το αναγνωρίζετε όλοι όσοι είστε νομικοί εδώ πέρα, ε, αν δεν είχαμε, θα ήταν πιο δύσκολο μάλλον αν δεν είχαμε σαφή νομική βάση. Αλλά και πάλι δεν αρκεί η νομική βάση. χρειαζόμαστε πολιτική βούληση, πολιτική συνεισφορά, ειδικά από τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι σήμερα είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε αυτό το στόχο. Γιατί ξέρετε ε, από τις μελέτες σας, τις σπουδές σας, ε, ότι σε καιρούς σαν σε καιρούς κρίσης, Συνήθως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση βρήκε τους πόρους και τη δύναμη να δράσει και να προχωρήσει προς τα μπρος στο ευρωπαϊκό αυτό πρόταγμα. Κυρίες και κύριοι, πέρα από τις ε, παρόλες τις βελτιώσεις που θα βρει κανείς ε, στη συνθήκη της Λισαβόνης, η καιρή είναι δύσκολη και για την Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαστε στη μέση μιας ιστορικής πρόκλησης. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τον, τον φόβο που αισθάνονται οι πολίτες ε, λόγω δύσκολων οικονομικών καιρών ένα φόβο που μπορεί να οδηγήσει εσωστρέφεια. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτούς τους καιρούς υπάρχουν, σε τέτοιους καιρούς υπάρχουν και ευκαιρίες. Ευκαιρίες για λαϊκισμό, ξενοφοβία, σοβινισμό, ε, και στο παρελθόν ε, συνέβησαν τα, ε, συνέβη κάτι τέτοιο και μπορεί να συμβεί και τώρα. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε αυτή την ηγεσία σε όλα τα ε, επίπεδα που να υποστηρίξει την Ευρώπη με λογικό τρόπο για όλους. Εγώ έκανα μια παρουσίαση κάποιων νέων εργαλείων καθώς και τις ευκαιρίες που, και τις προκλήσεις που βλέπουμε για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Υπάρχουν και εξωτερικά θέματα που αντιμετωπίζουμε. Σε... Ξέρω ότι σε αυτή τη συνδιάσκεψη θα αναπτυχθούν κάποια τέτοια θέματα. Ένα είναι σαφές. Με τη χρήση των εργαλείων που έχουμε για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, έχουμε μπροστά μας μια συνεχή διανοητική προσπάθεια. Πρέπει να δούμε τα γεγονότα, να τα ερμηνεύσουμε με καινοτόμο τρόπο και να βρούμε επικοδομητικές λύσεις για τις μελλοντικέ πολιτικές. Ελπίζω ότι θα αποφέρουν, αποφέρει πολλά ε, το, η συνδιάσκεψη Ζωμονέ με όλους εσάς και είμαι πεπισμένος ότι ε, θα βρούμε τρόπους να καλύψουμε τις προκλήσεις, θα κάνουμε χρήση των δυνατοτήτων, θα πρέπει να βρούμε και τα νέα εργαλεία, αλλά χρειαζόμαστε σαφώς νέα μέσα, νέες ιδέες, καινοτόμες. Είμαστε σε μια πορεία όπου αυτή η μάχη των ιδεών γιατί σε μάχη ιδεών βρισκόμαστε, έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Κατά τη δική μου άποψη, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αν δεν προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να οπισθοδρομήσει για πάντα. Έτσι τα βλέπουμε εμείς. Δεν είναι ε, να προχωράς επειδή είσαι πάνω στο ποδήλατο. Ε, ναι, από θεσμική απόψεω υπάρχουν πολλά τα οποία είναι απαραίτητα, αλλά δεν εννοώ αυτό. Με τις συνθήκες μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Υπάρχουν όμως κάποιες κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης όπου χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων αυτών που θα μας δώσουν νέες ιδέες. Η πρόσφατη αυτή κρίση μας καλεί να λάβουμε γρήγορα και ε, έκτακτα μέτρα. Ξέρετε ότι χρειαζόμαστε μια πιο δομημένη ευρωπαϊκή απόκριση. Τώρα, ε, πρέπει να ακούσουμε επίσης και τις κριτικές και να απορρίψουμε βέβαια τον επαγγελ... την επαγγελματική απεσιοδοξία σας. Μίλησα πιο πριν ε, για την ε, διανοητική ε, ζωφερότητα της απεσιοδοξίας, αυτό που λέμε τις κασάνδρες. Υπάρχει μια αγγλόφωνη, αν θέλετε, βιβλιογραφία για το ευρώ που θα έλεγα ευσεβείς ε, ε, πόθη, διότι περίμεναν να αποτύχει το ευρώ. Όχι, η δική μου ανάλυση είναι ότι το ευρώ θα πετύχει. Και θα πετύχει γιατί υπάρχουν βαθιά συμφέροντα στην οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης που απαιτούν την επιτυχία του. Πέρα από τη σπουδαιότητα του πολιτικού προγράμματος. Γι' αυτό το λόγο είμαι ότι η, ε, ευρώ, ε, το, το ευρώ είναι βασικό προσόν ε, και πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αν είμαστε όλοι μαζί, χωρίς να χάνουμε από τον ορίζοντα τις αξίες που μας ένωσαν πάνω από 50 χρόνια και που είναι περισσότερο σημαντικές από ποτέ. Και όπως είπα, έχετε σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, έχετε τη γνώση, την ανεξαρτησία, να βοηθήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δύσκολο καθήκον που την περιμένει. Και αυτό αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους υποστηρίζουμε αυτό το πρόγραμμα Jean και μάλιστα ε, στα επόμενα χρόνια σκοπεύουμε να το ενισχύσουμε και να το εδραιώσουμε, κυρίες και κύριοι. Η φετινή ε, συνδιάσκεψη έχει μαζέψει ε, πολιτικούς και διανοητές των πολιτικών θεμάτων. Πιστεύω ότι θα συζητηθούν πολλά σημαντικά θέματα τις επόμενες δύο μέρες, αλλά και η συμμετοχή τόσο πολλών ακαδημαϊκών δείχνει πόσο ελκυστικό είναι το πρόγραμμα Ζωμονέ και είναι αναγνώριση της ζωτικότητας της εμπειρογνωμοσύνης σας στον παγκόσμιο κόσμο, στην παγκοσμιότητα. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των προκλήσεων που έχουν τεθεί και το μόνο που μου μένει να κάνω είναι να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστώ για την προσοχή. Mr. President, thank you very, very much. Uh, you will not be able to uh, attend yourself uh, most of the discussion that is going to take place in this room today and tomorrow. But... Όλες, δυστυχώς δεν είστε σε θέση να παρακολουθήσετε όλες τις συζητήσεις βεβαίως, αλλά βεβαίως και θα σας ενημερώσουμε για την πρόοδο των εργασιών μας. Πιστεύω ότι οι καθηγητές μας συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τις θέσεις της Κομισιόν, κάποιοι τις αμφισβητούν τις θέσεις της Κομισιόν. Είμαι σίγουρος πάντως ότι θα γίνει έντονη και επικοδομητική συζήτηση, που σαφώς και θα βοηθήσει την Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε και πάλι Πρόεδρε. Τώρα, Έχουμε μαζί μας την κυρία Ντόρι Πακ, που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι τη γνωρίζουμε την κυρία Πακ, είναι από τα πλέον εξέχοντα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου έχει ήδη ε, επανειλημμένως βραβευθεί για το έργο της στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Εργάζεται σκληρά για την πρόθεση αυτών των ζητημάτων. Είναι πραγματικά προνόμιο να σας έχουμε μαζί μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μιλάω, θα μιλήσω γερμανικά. Uh, η γερμανική γλώσσα είναι μια πολύ ωραία γλώσσα και η μελωδία της χαράς ήταν ε, ούτως ή άλλως γερμανική όταν ε, ε, την συνέθεσε ο Μπετόβεν. Σε αυτέ... Εγώ δεν πρόκειται να κινηθώ βέβαια στα ύψη στα οποία μίλησε ο πρόεδρος. Εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, δουλεύω στο Κοινοβούλιο εδώ και 21 χρόνια. Έχω υπάρξει εισηγήτρια για την διαβίου μάθηση και στον τομέα της ε, και έχω υπάρξει εισηγήτρια για τον τομέα της εκπαίδευσης από την συνθήκη του Μάστριχτ. Χαίρομαι που μπορώ να λάβω το λόγο εδώ, που μπορώ να εκπροσωπήσω το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι το πρόγραμμα «ΖΩΜΟΝΕ» δείχνει όντως ότι έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία και ποια είναι η προσθέμενη αξία που μπορούν να δημιουργήσουν ε, τα ε, ευρωπαϊκά μέσα. Χαίρομαι λοιπόν που βλέπω τόσους ε, συναγωνιστέ σε αυτές τις ευρωπαϊκές ιδέες. Το θέμα μας σήμερα ονομάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν για όσα άλλαξαν για το Κοινοβούλιο, ήδη κάποια τα ανέφερε ο πρόεδρος της Κομισιόν και κάποια από αυτά που δεν ανέφερε ο πρόεδρο τη Κομισιόν, αλλά παρουσίασε, τη στρατηγική δηλαδή για το 2020, πώ αυτή θα λειτουργήσει στα δικά μας πλαίσια του Κοινοβουλίου. Η συνθήκη της Λισαβόνα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο σημαντικοί πυλώνες αλλά δεν, έχουμε, δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για όλα τα αποτελέσματα. Το πλεονέκτημα τώρα του Κοινοβουλίου πρέπει να πω ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας η, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται πιο διαφανείς και πιο δημοκρατικοί. Αυτό ήταν, αυτή ήταν πάντα η βασική μας θέση και από τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν ε, στην συνέλευση. Οπότε το ποτήρι είναι μισογεμάτο. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι καλύτερα, σαφώ. Αλλά νομίζω ότι προ το παρόν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που μα δίνει, με αυτά τα νέα, τι νέε ελευθερίε που μα δίνει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Καταρχήν, η συνθήκη τη Λισαβόνα δημιουργεί ένα πιο ε, ισχυρό νομοθέτη στο πρόσωπο του Κοινοβουλίου. Σε 40 επιπλέον τομεί πολιτική και καθώς επίσης και σε συνήθεις διαδικασίες όπως αυτή της συναπόφασης. Στους, ε, σε αυτούς τους, του, τους τομείς πολιτικής ανήκει και η γεωργία, η ενέργεια, η μετανάστευση, τα εσωτερικά, η, τα διαφορετικά ταμεία, η δικαιοσύνη και συνολικά μα υπάρχουν 86 νομικές βάσεις σε αυτή τη ε, διαδικασία. Και εκτός αυτού υπάρχουν και κάποιοι τομείς πολιτικής οι οποίοι δεν εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, στην υγεία, στην ενέργεια και επίσης στον αθλητισμό. Αλλά ξέρουμε ότι σχεδόν όλα όσα με τα οποία ασχολούμαστε εμείς στην Επιτροπή στην οποία είμαστε, είμαι πρόεδρος εμπίπτουν στον τομέα της επικουρικότητας, ακόμη και ο αθλητισμός. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο ήθελε φυσικά καλύτερο δημοκρατικό έλεγχο και ευθύνη λογοδοσίας. Και γι' αυτό θα ήθελα να... Και γι' αυτό μπορέσαμε και να ε, εκλέξουμε τον ε, νέο πρόεδρο της ε, Κομισιόν και τους εκπροσώπους και την εκπρόσωπο μάλλον για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Όλα αυτά για να γίνουν χρειαζόντουσαν την σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Αυτό αυξάνει και την νομιμοποίηση, τη δημοκρατική νομιμοποίηση για την οποία συνέχεια μην συζητούμε σήμερα. Πρέπει βέβαια ίσως ε, να κάνουμε πιο πολλές εκδηλώσεις ε, με τους, ε, με τους δημοσιογράφους ώστε να δούνε πόσο δημοκρατικό είναι το κοινοβούλιο Πολλέ φορέ η ε, ομάδα μας εδώ μας κατηγορείται ότι ε, είτε προσπαθεί να ενισχύσει την γερμανική κυβέρνηση είτε ότι προσπαθεί να τη ρίξει. Προσπαθούμε λοιπόν ε, να εκπονήσουμε πολιτική και να κάνουμε πολιτική υπεύθυνα για την Ευρώπη και χαίρομαι που είμαι εδώ και δεν βρίσκομαι πλέον στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Πιο πριν να μας είπε ο πρόεδρος Μπαρόζο ότι υπάρχουν επιπλέον αρμοδιότητες και σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συμφωνίες. Αυτό δεν είναι και πολύ ικανοποιητικό για κάποιες κυβερνήσεις. Σήμερα λοιπόν μιλούμε για διεθνείς συμφωνίες με τις οποίες, τις οποίες συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέες διαδικασίες ε, μετά τη θέση ισχύ της ε, συμφωνίας, της ε, συνθήκης συγγνώμη, οι οποίες προς το παρόν βρίσκονται σε φάση δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κομισιόν του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αλλά και εδώ θεωρώ ότι θα υπάρξει ε, αρκετός ε, έλεγχος από πλευράς Κοινοβουλίου. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την εκπόνηση του ε, προπολογισμού, το Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο. Γιατί η, η κατανομή σε υποχρεωτικέ και μη υποχρεωτικέ δαπάνε έχει καταργηθεί. Το Κοινοβούλιο θεωρείται ίσο λοιπόν με το Συμβούλιο των Υπουργών για όλο τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο μπορεί να επηρεάσει κάποιες δαπάνες οι οποίες μέχρι τώρα ήταν στην απληστική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι το Κοινοβούλιο στην απόφαση για την πολιετή χρηματοδότηση είναι, παραμένει πολύ περιορισμένο. Υπάρχει συμφωνία, αλλά δεν υπάρχει, ζητεί δηλαδή αλλά δεν υπάρχει συναπόφαση. Και στις τελευταίες δημοσιονομικές προοπτικές και ε, στι διαπραγματεύσεις η Επιτροπή του Κοινοβουλίου ε, έδρασε πολύ αποφασιστικά έτσι ώστε τα ε, κονδύλια για τον πολιτισμό και για την εκπαίδευση να αυξηθούν. Ανάγκασε λοιπόν το το, κοινοβούλιο, το Συμβούλιο να σταθεί στο ύψο των υποσχέσεών του. Εντάξει, δεν μα έδωσαν δισεκατομμύρια, αλλά εν πάση περιπτώσει μα έδωσαν κάποια εκατομμύρια παραπάνω. Και αυτό ε, πήγε, όλα αυτά τα επιπλέον κονδύλια πήγανε στον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Και αυτό πραγματικά με χαροποίησε πάρα πολύ γιατί ε, το έκανε η Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Πριν από 15 χρόνια δεν θα ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Χαίρομαι λοιπόν ε, και για τους ε, συναδέλφους από το Κοινοβούλιο οι οποίοι ε, και μέσω των εκλογικών τους περιφερειών ε, μου είπαν ότι όντω αυτός ο τομέας είναι πολύ σημαντικό, για τον οποίο πρέπει κανείς να έχει τα λεφτά στο χέρι. Οπότε στις επόμενες προοπτικές πρέπει να πω ότι και πάλι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, θα σηκώσουμε γη και ουρανό για να μπορέσουμε να αποφύγουμε να μας δώσουν λίγα ή λιγότερα χρήματα από ό,τι μας έδωσαν τώρα. Έχουμε λοιπόν επιπλέον δυνατότητα επιρροής μέσω της, συνθήκη μέσω της ε, συνθήκης της αλλά αυτό δεν είναι αυτός σκοπός. Δηλαδή δεν α, ε, ε, είμαστε εδώ εμείς οι, αυτοί που μπορούν να παίξουν τους κακούς και να λένε συνέχεια όχι. Σα θυμίζω ότι στην ε, συμφωνία σου είχαμε πει όχι. Και για σωστού λόγους είχαμε πει όχι. Και γι' αυτό τώρα έχουμε τη δυνατότητα, ναι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα, με τους Αμερικανούς να διαπραγματευτεί ένα νέο πακέτο ώστε να εξασφαλίσει την ε, ε, ασφάλεια των δεδομένων. Τώρα, έρχομαι στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 και της σχετικής στρατηγικής η οποία αναφέρθηκε από τον πρόεδρο της Κομισιόν. Τον Μάρτι παρουσιάστηκε η στρατηγική αυτή για τα επόμενα δέκα χρόνια. Θα ισχύει. Και θα σας θυμίσω ότι μιλούμε, υπήρχε και μια διαφορετική προσέγγιση δεν είχαμε προχωρήσει βέβαια τόσο την προηγούμενη φορά που συζητάγαμε το θέμα αυτό όσο θα έπρεπε, γιατί πραγματικά θεωρούσαμε ότι έπρεπε να επιτύχουμε τους ε, στόχους μας. Οι ουτοπίες και το να ευχόμαστε τα πάντα και τα οράματα, εντάξει είναι καλά, αλλά το πρόβλημα με την στρατηγική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 είναι ότι η Κομισιόν έθεσε κάποιους στόχους, ξέρει πού μπορούμε να αλλάξουμε κάτι και πού μπορούμε να πιέσουμε, αλλά όπως είπε ο πρόεδρο Μπαρόζο, φυσικά οι εθνικές κυβερνήσεις προσπαθούν συνέχεια να ζητήσουν κάτι παραπάνω, να μας ζητήσουν χρήματα, κονδύλια στο χέρι, γιατί πρέπει να απόσχουν από κάποιε δραστηριότητε. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θα προσπαθήσει να εξισορροπήσει τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με τη στρατηγική αυτή. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να σα πω, οι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο είναι απολύτως, ε, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι για το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί γιατί δεν γίνεται μέσα μια στρατηγική μέχρι το που θα ισχύει μέχρι το 2020 έτσι να, το, να τις δώσουμε τις ευλογίες μας ε, ρίπη οφθαλμού. Με την, ε, θέλουμε να έχουμε λόγο σε όλη αυτή τη διαδικασία, στην εκπόνηση, στην εξέλιξη αυτή τη διαδικασία ώστε να επιτύχουμε του ε, στόχου και ούτω ή άλλω είμαστε και συνυπεύθυνοι γι' αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μεγαλύτερο χρόνο. Η Κομισιόν σωστά έδωσε μια πολύ κεντρική σημασία στην όλη αυτή διαδικασία η Κομισιόν για την καινοτομία, την κινητικότητα, την έρευνα και την εκπαίδευση. Όλοι αυτοί είναι τομεί στους οποίους εμείς μόνο εν μέρη είμαστε υπεύθυνοι και μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε. Κάποιοι τομεί, όπως σας είπα, ήδη εμπίπτουν στον τομέα τη επικουρικότητα. Γι' αυτό ε, και, το, και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν από κοινού πρέπει να προχωρήσουν στους τομείς αυτούς γιατί θεωρούμε ότι όταν προχωρούμε από κοινού μπορούμε να έχουμε περισσότερες ε, δυνατότητες να πείσουμε και τις κυβερνήσεις. Στους τομείς λοιπόν αυτούς υπάρχουν κάποιες ναυαρχίδες, έτσι τις λέμε. Και μια ναυαρχίδα είναι Youth on, είναι το Youth on the Move, οι νέοι δηλαδή, η κινητικότητα των νέων. Ελπίζω να μπορέσουμε να, την, ε, να, δώσουμε περισσότερη ζωή σε αυτή την ε, σε, αυτή την, ε, σε αυτόν τον τομέα, σε αυτή την Έχουμε τώρα μια αυαρχίδα που αφορά τους νέους. Εμείς είμαστε μια γυράσκουσα κοινωνία. Και μιλούμε τώρα εδώ για την διαβίου μάθηση, την οποία δεν θέλουμε να δώσουμε, στην οποία δεν θέλουμε να δώσουμε τη σημασία που πρέπει. Η διαβίου μάθηση είναι πολύ σημαντική αυαρχίδα για τη δική μας την δουλειά. Γι' αυτό υπάρχει ο Λεωνάρντο, γι' αυτό υπάρχει το Ζαρμονέ, γι' αυτό υπάρχει ο Γκρούντβιχ, γι' αυτό υπάρχει ο Κομένιος, γι' αυτό υπάρχει ο Εράσμου. Υπάρχουν πολλοί τομεί οι οποίοι δεν θεωρούνται κατά ανάγκη, δεν εμπίπτουν κατά ανάγκη στα πλαίσια του Youth on the Move. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω την Κομισιόν. Εγκάρδια, ούτω ή άλλω δική τη ιδέα ήταν και στο παρελθόν το λέγαμε. Δεν θέλω να σα φάω τη δόξα, αλλά θα ήθελα να μην μας δυσκολέψει η Επίτροπος για την εκπαίδευση. Αυτό το Youth on the Move πρέπει να το εφαρμόσετε ένα προς ένα. Youth on the Move μπορεί να, φορά τις, μπορεί να, μπορεί να αντικαταστήσει το, ε, τα προγράμματα για τους, ε, για τους νέους. Μπορεί όμως να έχει επίδραση και στη διαβίωμάθηση. Σας παρακαλώ λοιπόν, σας παρακαλώ πραγματικά αφήστε τη διαβίου μάθηση ως μεμονωμένη, ε, μεμονωμένο τομέα. Δημιουργήστε την ε, διαβίου μάθηση και μπορούμε να δημιουργήσουμε εξαιρετικές συνέργειες με αυτό. Σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα εδώ γιατί ήδη τα έχω πει εγώ και στην Επίτροπο και σε άλλους, αλλά Ελπίζω ότι σήμερα έτσι με το επίσημο αυτό αίτημά μου που δεν το κάνω μόνο ως Τόρις Πάγκ αλλά και ως ε, ε πρόεδρος της Επιτροπής ελπίζω να σας έχω πείσει και οι συναδελφοί μου λένε ότι χρειαζόμαστε μία μεμονωμέ... ένα μεμονωμένο τομέα για τη διαβίου μάθηση και πραγματικά θα ήθελα την υποστήριξή σας. Κυρίες και κύριοι, σας είπα η διαβίου μάθηση είναι σημαντική για μας και για την πολιτική εκπαίδευση και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στα τελευταία χρόνια και από την Κομισιόν και θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω και τον κύριο Κεντάν που ήταν ο ε, προκάτοχος του κυρίου Τρουσίνσκι ε, ότι μας έχει φέρει σε σημείο να σκεφτούμε, να δούμε πώς μπορούμε να συγκρίνουμε τα συστήματά μας. Είναι απαραίτητο αυτό. Δεν θέλουμε να καταργήσουμε κάτι, δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε στους ανθρώπους να συμμετάσχουν, αλλά θέλουμε να συμμετάσχουμε με το μεγαλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό πάντα το έλεγε η Κομισιόν και αυτό το θεωρώ καλό. Οπότε, σε σχέση με αυτό, να πω και το εξή. Ελπίζω η νέα πολιτική και το νέο πρόγραμμα για τη διαβίου μάθηση να έχει έναν τομέα στο Κομένιους που να ονομάζεται Comenius Teacher, δάσκαλοι. Χρειαζόμαστε καλύτερους δασκάλους, καλύτερους καθηγητές, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στα σχολεία. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν ε, δάσκαλοι ή καθηγητέ που δεν έχουν ιδέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν ε, ενδιαφέρονται καν. Πολλό δε μάλλον να ε, κινητοποιήσουν και τα παιδιά του που έχουν στι τάξει του να ενδιαφερθούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν στα πλαίσια του προγράμματο για τη διαβίου μάθηση θα πρέπει να υπάρξει ένα τμήμα που να αφορά του καθηγητέ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Κυρίε και κύριοι, η πολιτική βούληση όμω πρέπει να υπάρχει ούτω ή άλλω πέρα από τα κονδύλια γιατί αλλιώς ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά που θέλουμε. Γι' αυτό με τις, στις επόμενες ε, δημοσιονομικές προπτικές ε, θα, αγωνιστούμε γι' αυτό ώστε η επόμενη γενιά τα... το να μπορεί να υποφεληθεί του πολίτους προγράμματος για την εκπαίδευση και το πρόγραμμα αυτό να λάβει περισσότερα κονδύλια. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το πόσο, πόσο σημασία δίνουμε στην πρόθεση των τομέων αυτών, γιατί μιλούμε συνέχεια για την κρίση. Η κρίση αυτή μπορεί να λυθεί μόνο εάν ενισχύσουμε αυτούς τους τομείς. Και σας παρακαλώ, όπου και να είμαστε, αυτό ακριβώς να ζητούμε. Παντού. Πρέπει να έχουμε πιστικά επιχειρήματα και αυτά τα έχετε ούτως ή άλλως όλοι. Καταρχήν, τα προγράμματα που ανήκουν στην, στον τομέα της παιδείας αποτελούν τα πιο επιτυχή προγράμματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Εράσμους, το Κομένιος, ο Γκρούντβιχ, ο Λεωνάρντο, Όλα αυτά είναι, και το Ζαμονέ βεβαίω, είναι προγράμματα που πραγματικά έχουν μεγάλη επιτυχία. Είμαστε, είναι πολύ δημοφιλή. Το πρόβλημα λοιπόν της ροής των κονδυλίων δεν υπάρχει στα προγράμματα αυτά. Για πολλά προγράμματα υπάρχει, αλλά για αυτά δεν υπάρχει. Συνήθως έχουμε πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε να δώσουμε. Και αυτό αφορά τους ανθρώπους άμεσα. Δημιουργούμε ε, ορατότητα, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία. Έχουμε μια ανοιχτή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό βοηθούμε και την εκμάθηση γλωσσών, καθώς και άλλες, άλλα βασικά προσόντα. Τώρα, η αναγκαιότητα της, ε, το να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, σε διάφορες κοινωνίες, ε, οι οποίες ε, έχουν διαφοροποιημένες κοινωνίες, πιέζονται και από την παγκοσμιοποίηση, δεν μπορούμε να έχουμε 50% των μαθητών οι οποίοι να διακόπτουν τις σπουδές τους. Επίσης, παιδιά που, έχουν, που είναι μετανάστες ή παιδιά μεταναστών δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας. Τρίτον, όλα αυτά είναι επιχειρήματα που σας λέω. Η πολιτική εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ενισχύσει τις εθνικές πολιτικές παιδείας. Το έχω ξαναπεί αυτό. Το πρόγραμμα Εράσμους έχει πραγματικά, είναι αποφασιστική σημασία. Δυστυχώς, η διαδικασία της Μπολόνια δεν πήγε τόσο καλά δεν θέλω τώρα να πω σε λεπτομέρειε. Δεν είναι κάτι για το οποίο, το οποίο, το οποίο η Κομισιόν. Είναι κάτι το οποίο δεν προώθησαν πολλοί κυβερνήσεις, τα πανεπιστήμια. Εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ ότι αυτή η διαδικασία, που είναι πολύ σημαντική διαδικασία, θα έπρεπε να έχει συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ή τα εθνικά κοινοβούλια, αν το είχαν συζητήσει, αυτή η διαδικασία της Μπολόνια δεν θα είχε α, δομηθεί με τέτοιο με τσιλαθασμένο τρόπο. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους που σας είπα, πρέπει να έχουμε και, με, να έχουμε και άλλους εκτός από αυτούς για να μπορούμε να ζητούμε ε, παραπάνω κονδύλια. Να έχουμε λοιπόν ε, εναλλακτικέ. Πρέπει να σκεφτούμε, και το έχω πει πολλές φορές, ε, ελπίζω οι Γεωργοί να μην μου θυμώσουνε, αλλά έχουμε 880 εκατομμύρια ευρώ στην Γεωργία κάθε χρόνο ενώ έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο για όλα τα προγράμματα ε, ε, που αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στην, ε, στους ανθρώπους. Φυσικά οι επιτυχίες στον τομέα αυτό μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση σε εθνικό επίπεδο σε εθνικό επίπεδο δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την εθνική πολιτική εκπαίδευση. Μπορούμε να την ενισχύσουμε, μπορούμε να την προωθήσουμε για την ε, επαγγελματική εκπαίδευση, για τους, ε, για τον, ε, για τους νέους και για, την, για τον πολιτισμό. Υπάρχουν τέτοια μεμονωμένα προγράμματα. Ελπίζω σε αυτό να μπορέσουμε σε, αυτό το, σε αυτή την υπουργική διάσκεψη των Υπουργών παιδείας να τα συζητήσουμε όλα αυτά έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις αρνητικά, σχόλια, θετικά για να μπορέσουμε να μάθουμε ένας από τον άλλον. Περνάμε δύσκολες ώρες, οι επενδύσεις είναι όλο και, γίνονται όλο και πιο δύσκολες, πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους, στους νέους, αλλά και στους ε, μεγαλύτερους στην προώθηση της εκπαίδευσής τους, στην καινοτομία τους, στη δημιουργικότητά τους η οποία είναι ο καλύτερος μακροπρόθεσμα τρόπος ώστε η Ευρώπη να εξασφαλίσει το μέλλον για τους νέους της. Αυτή λοιπόν είναι η δική σας δουλειά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για την προσοχή σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Uh, uh, Ευχαριστούμε πολύ Κυρία Πακ, κυρία Πρόεδρε της ε, Επιτροπής Παιδείας και εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστούμε για την ε, τόσο σαφή παρουσίαση της εκπαιδευτική πόλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, Ιδίω σε συσχετισμό και με τη στρατηγική ΕΕ 2020. Με την ευκαιρία αυτή, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχαριστήσουμε θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την διοργάνωση της διάσκεψης αυτής στον οίκο σας. Βεβαίως ανέκαθεν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριζε στενά το πρόγραμμα Jean Monnet και τις διασκέψεις μας. Έχουμε μαζί μας πράγματι τον καθηγητή Χωσέ Μαρία Χιλ Ρόμπλες που αυτά αποδεικνύει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο καθηγητής ε, προεδρεύει της Ένωσης πρώην Ευρωβουλευτών και ταυτόχρονα προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Συμβουλίου για τη δράση Ζωαμονέ. Ευχαριστώ θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την φιλοξενία σας, τα χτίρια σας. Uh, uh, uh, να περάσουμε τώρα στα επόμενα μας σημεία. Πρόεδρε, παραμένετε μαζί μας. Να περάσουμε και σε κάτι πιο ευχάριστο. Πολλά φαίνεται ευχάριστα βεβαίως αυτή τη διάσκεψη. Απονομή του βραβείου Ζαμονέ για το 2010. Με χαρά μου θα δώσω το λόγο στο αφεντικό μου, στην Επίτροπο Αντρούλα Βασιλείου που έχει την αρμοδιότητα στο πλαίσιο της Κομισιόν για την παιδεία εκπαίδευση, την πολυγλωσία και την νεότητα, η Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κυρία Πάκης και κύριοι, πρώτα απ' όλα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας και την ε, κυρία Ντόρι Πακ διότι μας αφιερώνουν χρόνο από τον τόσο του πολύτιμο χρόνο ε, πράγματι ήταν προνόμιο για όλους μας ε, το γεγονός ε, ότι συνεισφέρετε με τα φώτα σας σε αυτές τις εξελίξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι για μένα η πρώτη μου τέτοια διάσκεψη ε, υπό την αρμοδιότητα πλέον ε, της Επιτρόπου για θέματα παιδείας, εκπαίδευσης, αθλητισμού, νεότητας και πολυγλωσίας. Είναι υπέροχο το ότι αναλαμβάνω πρωταγωνιστικό ρόλο ε, στο ευρωπαϊκό μέτωπο για τέτοια θέματα που άμεσα επηρεάζουν τη ζωή, τη ζωή του Ευρωπαίου πολίτου. Και είναι και μεγάλο προνόμιο που έχω την αρμοδιότητα για το πρόγραμμα Jean Monnet, όπως μας έχουν αποδείξει προσφάτες εξελίξεις, αμφισβήτητα, το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την περαιτέρω ενοποίηση με βάση την ευθύνη και την αλληλεγγύη. Για να επιτύχουμε θα πρέπει να αναλυφθεί δράση σε τεκμηριωμένη βάση, σωστό προβληματισμό και διανοητική συνεισφορά. να, να δούμε αυτή τη διάσκεψη των καθηγητών Ζαμονέ. Monnet. Εσείς, και αν έχετε την πραγματογνωμοσύνη και το κριτικό πνεύμα, και την αξιοπιστία και εκπροσωπούνται ε, τους πλέον εξέχοντες Διανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδού περίτρανα η πιο, ε, ιδού η απόδειξη της αξίας του Ζαμονέ. Αλλά τώρα πλέον θα περάσουμε στην απονομή του βραβείου Ζαμονέ 2010. Όπως γνωρίζετε το, θε, το, η διαβίου μάθηση απονέμει κάποια βραβεία για να βραβεύσει την αριστεία κατά την εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων. Οπότε αποφασίσαμε να συνεχίσουμε αυτή την πρακτική και να προχωρήσουμε σε απονομή ενός βραβείου Jean Monnet το χρόνο στην ετήσια διάσκεψη Jean Monnet. Όπως κάναμε και τις προηγούμενες χρονιές, η επιλογή πράγματι έγινε υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Χωσέ, Μαρία Χίλ Ρόμπλες, που είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Συμβουλίου για το πρόγραμμα Jean Monnet, και του καθηγητή Αρίκε Μπανούς που είναι ο πρόεδρος του Παγκοσμίου ECSA. Θα ήθελα να καλέσω και τους δύο κυρίους να πάρουν το λόγο για να μας πούν δύο λόγια σε σχέση με το πρόγραμμα Jean Monnet και το βραβείο. Θέλουμε να κρατήσουμε όμως το σας μέχρι το τέλος. Ε? Μην αποκαλύψετε το παραμικρό, κύριε καθηγητά. Ο καθηγητής ε, Χωσέ Μαρία Χιλερόμπλες. Ευχαριστώ Επίτροπε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας στο βραβείο αυτό και εν γέννη στη δράση Ζαμονέ. Εξ ονόματος ολίκληρης της κοινότητας Ζαμονέ να σας πω ότι είμαστε κατευχαριστημένοι με το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Κομισιόν εξήγηλε τον δικό σας διορισμό σε θέματα πολυγλωσίας, εκπαίδευσης, παιδείας, νεότητας και αθλητισμού. Πράγματι θέλουμε μια εξέχουσα προσωπικότητα ε, σε θέματα παιδείας και νομίζω ότι χάρη σε εσά είναι λαμπρό το μέλλον που μας περιμένει. Βεβαίω και χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια. Είμαστε βέβαιοι ότι θα πάει να τα διεκδικήσει η Ντόρις, εξ όλων μα από το 89 που άρχισα να πρωτοεργάζομαι στην Επιτροπή Παιδεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τότε τα διεκδικεί αυτά τα κονδύλια η Doris και, πακ ε, και πολύ χαίρομαι που συνεχίζει να τα διεκδικεί. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, Πρόεδρε, να σα ευχαριστήσω όλο ιδιαίτερος για τη στήριξή σα και για τη συμβολή σας Βλέπ, χαίρομαι με το ζήλο σας. Πράγματι θέλετε η Κομισιόν τις τόσο αυτές λεπτές στιγμές να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Είναι απαραίτητος ο ρόλος αυτός της Κομισιόν. Δεν φτάνει η διακυβερνητική και μόνο διευθέτηση στο πλαίσιο της νέας οικονομικής διακυβέρνησης. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι ε, επιμένει, εμένει στο ρόλο της η Κομισιόν. Και ορθά το έχετε τονίσει κι εσείς, είναι απαραίτητος ο κοινοβουλευτικός έλεγχος εφόλης της διαδικασίας. Είναι κέρια σημασία αυτό. Το έχω σημειώσει προσεκτικά. Την ερχόμενη Δευτέρα, όταν στη Μαδρίτη θα απευθυνθώ στο Συμβούλιο μας για θέματα συνεργασίας μεταξύ ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων για θέματα που αποτελούν απόρρια της ηθίκης της Λισαβόνας, το κλειδί είναι πώς πετυχαίνουμε την πιο αποτελεσματική συνεργασία με την Κομισιόν σε θέματα οικονομικής, ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. βαθμιαία δείχνεται όλο και μεγαλύτερο ζήλο σε, σε αυτό το δίκτυο παρά τη βαρυφορτωμένη σας ατζέντα έρχεστε και είστε παρόν μαζί μας στην ετήσια μας διάσκεψη. Κάθε χρόνο αυτό βλέπουμε. Βεβαίω και οι καθηγητέ μα, ε, οι καθηγητέ Ζωαμονέ είναι πάντα στη διάθεσή σα. Είναι πρόθυμοι πάντα να σα στηρίξουν. Θα ήθελα βεβαίω να χαιρετήσω και την συνάδελφο κυρία Πακ. Τόσα χρόνια δουλέψαμε μαζί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε φίλοι. Η Τόρις έχει μεγάλο δυναμισμό, δείχνει τεράστιο ζήλο στα θέματά μας και αυτό εδώ και χρόνια. Ε. Και ακόμα και σήμερα το πρωί το είδαμε από την ομιλία σας με τις διεκδικήσεις σας και το δυναμισμό σας. Είναι τυχερή η παιδεία στην Ευρώπη που σας έχει στην Προεδρία της Αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε που είμαστε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε για την σημερινή φιλοξενία, ιδού η απτή απόδειξη της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκού κόσμου, Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόεδρε Μπαρόσο, Επίτροπε Βασιλείου, κυρία Μπάκε, Πάκε. Αυτή την τόσο λεπτή στιγμή για την Ευρώπη τώρα είναι που χρειάζεται καλύτερη κατανόηση θεμάτων ευρωπαϊκής ενοποίησης σε καθημερινή, ε, ε, και ολοκλήρωση σε καθημερινή βάση. Το μήνυμά μου είναι το εξή, ότι η κοινότητα Ζαμονέ είναι έτοιμη να αναλάβει τι ευθύνε τη και να παίξει το δικό τη ρόλο. Είμαστε εντελώ αποκεντρωμένοι. Έχουμε κέντρα και έδρες ε, σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης και παραπέρα. Μιλάμε για απόλυτη αυτονομία, ε, με πνεύμα, άρα το δίκτυο Ζαμονέ είναι από τα πλέον αξιόπιστα μέσα για να καλυφθεί το χάσμα της γνώσης σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά θέλω να τονίσω. Αυτονομία και κριτικό πνεύμα. Διότι αυτός είναι ο κύριος ρόλος των καθηγητών Ζαμονέ. Να πάνε να εξηγήσουν τι εστί ευρωπαϊκή πολιτική και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι απαραίτητο το έργο τους. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα βεβαίως έχουν και άλλα μέσα για σωστή ενημέρωση για σωστή διαπαιδαγώγηση. Το πρόγραμμα Jean Monnet έχει τη δική του συγκεκριμένη αποστολή. Ο ρόλος μας είναι πολύ συγκεκριμένος. Εξηγούμε την όλη ιστορική διαδικασία και τις διάφορες τις φάσεις. Επεξηγούμε τους λόγους πίσω από την κάθε φάση ακολουθώντας καθαρά επιστημονική προσέγγιση. Προσέγγιση που διαφέρει ανάλογα με το που βρίσκεται η έδρα. Αν βρίσκεται στην Ευρώπη, στην Ασία, στη Βόρεια Αμερική, στην Νότια Αμερική, στην Λατινική Αμερική, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία. Και προφανώς οι προσδοκίες αναπεριφέρουν διαφορετικές. Το παν είναι οι μαθητές να διδαχθούν ε, κάποια κλειδιά για να αντιληφθούν κάποια πράγματα και να παρακολουθούν πιο εύκολα. Υπάρχουν και κάποια χέγγια σε αυτή τη ε, διαδικασία βεβαίως και έτσι ε, φέρνουμε εις πέρα στην αποστολή μας. Την αποστολή της διαπαιδαγώγησης. Το δίκτυο Jean Monnet θα πρέπει ε, βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κομισιόν και αυτή ήταν η ορθή απόφαση. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με μία πρόταση. Είναι εκατοντάδες τα κέντρα αριστείας, Ζωμονέ, ανά τον κόσμο. Μιλάμε για πανεπιστήμια σε 62 χώρες και στις 5 υπήρους. Το δίκτυό μας καλύπτει κάθε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρα είναι πραγματική πηγή το δίκτυό μας και όντως μπορεί να σας παρέχει αξιόπιστες συμβουλές για τη χάραξη πολιτικής. Και στρέφομαι και προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαρίστως να σας παρέχουμε την πραγματογνωμοσύνη μας. Ιδίω σε συσχετισμό με τη στρατηγική ΕΕ 2020 και παραπέρα και ευχαρίστω να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σα. Είναι μεγάλη η πραγματογνωμοσύνη των καθηγητών μα. Πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε επικοδομητικό ρόλο. Μπορούμε να σας στηρίξουμε χάρη στην αυτόνομη μας ανάλυση και παροχή συμβουλών για θέματα επικαιρότητα άμεσα και αμερόληπτα και ανιδιοτελώς. Ευχαρίστως σε συσχετισμό με τη στρατηγική ΕΕ 2020 και πάρα να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Είμαι πεπισμένος ότι στο νέο νομοθετικό και στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε πολλά να προσφέρουμε. Είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε πάντοτε την υποστήριξή σας και οι σημερινές σας δηλώσεις αυτό άλλωστε αποδεικνύουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε καθηγητή Χιλ Ρόμπλες. Σας ευχαριστούμε για τον ζήλο σας στο πρόγραμμα Ζαμονέ. Ε, έχετε ένα εξαιρετικό υπόβαθρο ως πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέκαθεν ήσασταν σε ρόλο ευθύνη, εσεί και αν είστε ο καλύτερο πρέσβη για το πρόγραμμά μα. Σα ευχαριστούμε για την προσφορά σα να συμβάλλετε με κάθε τρόπο στο πλαίσιο τη στρατηγή ΕΕ 2020. Βεβαίω και θα τη δεχτούμε την προσφορά σα. Τώρα ο καθηγητή Μπανού έχει το λόγο που έχει την έδρα Ζαμονέ και είναι πρίτανης ε, ε, ανθρωπίνων επιστημών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας. Σήμερα βεβαίως βρίσκεται ανάμεσα μας ως πρόεδρος του Παγκοσμίου ECSA, που σημαίνει ότι εκπροσωπούνται ενώσει πανεπιστημιακές ενώσεις από 58 διαφορετικέ χώρες. Θα ευχαριστήσω και εσάς και τις εθνικέ E.C.S.A. για το εξαιρετικό σας έργο. Κύριε Καθηγητά. Ευχαριστώ, κυρία Βασιλεία. Και εκ ε, Ομοσπονδίας Σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, υποστήριξή σας. Χαίρομαι πολύ που από κοινού και με εσά και με τον Γενικό Διευθυντή του Σίνσκι ε, θα είμαστε ο συνομιλητής ε, για τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο Μπαρόσο που εδώ και χρόνια διατηρεί τον διάλογο μαζί μας και πιστεύω ότι θέλω να ευχαριστήσω μάλλον και την Doris Πακ για την ε, πραγματικά πολύ αποτελεσματική δουλειά που κάνει στην Επιτροπή ε, Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τιμή μας που έχουμε μια τόσο αποφασιστική φίλη, θα μπορούσα να πω, στο Κοινοβούλιο. Ποιοι είμαστε. Είμαστε εκπρόσωποι ακαδημαϊκών που, αφορούν, που ασχολούνται με, με ευρωπαϊκά θέματα ένα δίκτυο καθηγητών και ερευνητών για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενεργών σε 58 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα μέλη μας είναι ακαδημαϊκοί που ε, κάνουν ε, έρευνα, ε, που διδάσκουν και θέλουν να αυξήσουν την ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν ανεξάρτητο και δυναμικό τρόπο. Στα πλαίσια αυτά συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις που έγιναν από τον καθηγητή Χιλ Ρόμπλε για το μέλλον και την, ε, το συσχετισμό των Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Σπουδών. Να κάνω όμως και ένα επιπλέον σχόλιο για το μέλλον. Θυμάμαι ότι πριν από τη δημιουργία του προγράμματος για τη διαβίου μάθηση, κάποιος έλεγε ότι το πρόγραμμα μπορεί να ε, ενσωματωθεί στο πρόγραμμα το οποίο ε, με το οποίο ασχολείται η Γενική Διεύθυνση για την, για την Επικοινωνία. Η Κομισιόν, ε, υπό την Προεδρία του Πρόεδρου Μπαρόσου, έκανε σωστή επιλογή όταν πρότεινε το πρόγραμμα αυτό να ενσωματωθεί στο, στη νομική βάση ε, για την εκπαίδευση. Οι καθηγητές Ζαν Μονέ είναι ε, λέκτορες και ερευνητές, ανεξάρτητοι καθηγητές, δεν είμαστε λοιπόν ε, στον τομέα του να πουλήσουμε την ε, Ευρώπη. Ε, έχω λοιπόν πραγματικά μεγάλο, μεγάλο σεβασμό για την πολιτική επικοινωνία η οποία τόσο πολύ χρειάζεται. Μπορούμε λοιπόν, τα μέλη μας μπορούν να θέτουν ερωτήματα, να χρησιμοποιούν ή να ψάχνουν να βρουν επιχειρήματα και μερικές φορές να διαφωνούν κιόλας. Η δική μας δουλειά και το δικό μας πάθος είναι κριτικός να αναλύουμε την διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το critical e βέβαια το εννοώ με την καλή έννοια. Είμαστε η ενδιάμεση ε, σε ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα, το πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε η ενδιάμεση μεταξύ της ε, νέας γενιάς, προς τη νέα γενιά μάλλον, που θα αναλάβει την ευθύνη για το ευρωπαϊκό προ, για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και θα είναι και οι μελλοντικοί καθηγητέ. Το δικό μα καθήκον δεν είναι να πληροφορήσουμε, αλλά να μορφώσουμε, να δημιουργήσουμε αξιοπιστή ε, ε, αξιοπιστία, εμπιστοσύνη μέσω συγκεκριμένων επιχειρημάτων. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο σα υποβάλλω το ότι δεν μπορούμε να είμαστε τμήμα ενός ε, προγράμματος επικοινωνίας γιατί η δική μας φύση είναι πιο κοντά στα υπόλοιπα προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση και το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν περίπου 8.000 εμπειρογνώμονες που θέλουν να κάνουν διάλογο, να σκεφτούν, να συμβουλεύσουν. Ίσως είναι μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές σκέψεις στον κόσμο η δική μας. Και είμαστε πεπισμένοι ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι και πρέπει να είναι το υπόδειγμα από την Ευρώπη. Τώρα για το βραβείο Ζαμονέ. Από την διάσκεψη για την, ε, που ξεκίνησε την, ε, το πρόγραμμα Ζαμονέ υπάρχει αυτό το ετήσιο βραβείο για να βραβεύσει την αριστεία σε ευρωπαϊκές σπουδές κάθε χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τον καθηγητή Χίλ ρόμπλε ως Προέδρου του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το, πρόγραμμα, για το πρόγραμμα Ζαμονέ και από μένα ως ε, ε, πρόεδρο του Δικτύου να προτείνουμε μέλη για το δίκτυο Ζαμονέ, καθηγητές που είναι γενικώ αναγνωρίσιμοι για την αριστεία τους και για την ευρεία συμβολή τους στην ολοκλήρωση των ε, εκπαιδευτικών δομών και των δικτύων που έχουν, ε, που έχουν ε, άμεσες επιδράσεις στην διαβίου μάθηση. Στις 30 Απριλίου, μετά από πολλές ανταλλαγές και διαβουλεύσεις, τρία ονόματα υπευλήθησαν με σειρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, η τελική επιλογή ε, θα γίνει από την Επίτροπο, έγινε μάλλον από την Επίτροπο Βασιλείου. Οπότε δεν είμαι εγώ αυτός που θα πει και το βραβείο πάει στον ή στην. Σας ευχαριστώ. Well, ladies Κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, συνολικά η κοινότητα Ζωμονέ είναι ένα παράδειγμα ε, ακαδημαϊκής ε, αριστείας και δέσμευση στις μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως τα κριτήρια ξεπερνούν ε, τα ακαδημαϊκά κριτήρια για την απονομή των βραβείων 2010. Ε, επιλέξαμε να απονείμουμε τα βραβεία 2010 με βάση τον ε, πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισαν ε, αυτοί οι οποίοι κερδίζουν αυτά τα βραβεία της έδρας Ζωμονέ για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών σπουδών κατά τη δύσκολη μεταβατική περίοδο σε κάποιο από τα πρόσφατα κράτη-μέλη. Οπότε με χαρά ανακοινώνω ότι το βραβείο Ζωμονέ απονέμεται στον καθηγητή Τιμπορ Παλάνκαη Ο καθηγητής Παλάνκα είναι διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών και Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κορβίνου της Βουδαπέστης. Η δημιουργία των Ευρωπαϊκών Σπουδών στην Ουγγαρία ως αναγνωρισμένο πεδίο ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας οφείλει πολλά στον καθηγητή Παλάνκαη. Το 1993 όταν άνοιξε για πρώτη φορά η δράση Jean Monnet για αιτήσει ε, Ουγγρικών Πανεπιστημίων ε, του δόθηκε άμεσα η έδρα Ζωμονέ και μετά έδρα ad persona. Δεν είναι εκπληκτικό αυτό, δεν προκαλεί έκπληξη, διότι ε, ως πρωτεργάτη στον τομέα αυτό, ο καθηγητής Παλάνκαη δίδασκε πράγματα για την Ευρωπα... τις ευρωπαϊκές κοινότητες πριν από τη λήξη του ψυχρού πολέμου. Ως δυναμικός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής, της Ουγγρικής Ένωσης για τις, ευρωπαϊκές, ε, για τις ευρωπαϊκής κοινότητας, ο καθηγητής Παλάνκαη και το πρόγραμμα ζώμονε διαδραμάτισαν σημαντικότατο ρόλο για την επέκταση της διάδοση της διδασκαλίας της ευρωπαϊκής Ολοκλήρωση ε, ολοκλήρωσης σε όλα τα ουγγρικά πανεπιστήμια, σε όλα τα επίπεδα, από τις βασικές σπουδές μέχρι τις μεταπτυχιακές και τα διδακτορικά. Ε, ήδη από το 1990 τότε υπήρχαν μόνο μερικές, ε, μια δωδεκάδα περίπου ε, εμπειρογνώμονες στην Ουγγαρία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 250 καθηγητές και βοηθοί οι οποίοι συμμετέχουν στη διδασκαλία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στη χώρα. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι και οι καθηγητές από την Ουγγαρία ε, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ε, ενταξιακή διαδικασία, όπως και οι καθηγητές Ζων Μονέ σε πολλά άλλα κράτη-μέλη. Επ' αυτή την έννοια θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στα δυναμικά μέλη του δικτύου μας, στα νεότερα κράτη-μέλη. Καθηγητά Παλάνκα, είστε ένα εξέχον παράδειγμα της ε, ολόκληρης της κοινότητας Ζωμονέ. Παράλληλα δημιουργήσατε μια για γέφυρα ανάμεσα στις διαφορετικές διαστάσεις του προγράμματος Ζωμονέ. Επιπλέον ε, Εκτός από την έδρα σας Ζωμονέ στο Πανεπιστήμιο Κορβίνους, ε, διδάξατε για 10 χρόνια στο Κολέγιο της Ευρώπης, που είναι ένα άλλο, αν θέλετε, παρακλάδι της ε, ε, άλλο ένα ε, κόσμημα κατά κάποιο τρόπο, ένας άλλος πολύτιμος λίθος στο, στο στέμα του Ζωμόνα επιπλέον. Είστε μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Συμβουλίου για το πρόγραμμα Ζωμονέ και για όλους αυτούς τους λόγους ε, συμβολίζεται τη δέσμευση ε, στα ευρωπαϊκά προγράμματα και αυτό το βραβείο είναι ένα δείγμα της μεγάλης εκτίμησης που σας αποδίδει η ακαδημαϊκή κοινότητα. Well, Βεβαίως έχω συγκινηθεί βασίτατα και δεν μπορώ να πω τίποτα. Θα πρέπει να πω ότι η απόφαση για το πρόγραμμα Ζωμονέ ε, επεκτάθηκε ευθύς εξ αρχής στα νέα κράτη-μέλη και έχει ιστορική σημασία διότι μας βοήθησε να ξεκινήσουμε μαθήματα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για να βοηθήσουμε τα μέλη μας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ε, του μέλλοντος. Οπότε ε, είναι δύσκολο να υπερεκτιμήσει κανείς ε, την σπουδαιότητα του ζώμων. Θέλω να σας ευχαριστήσω και σε όλες τις γλώσσες, όχι μόνο στα γαλλικά το ευχαριστώ, αλλά και στα ουγγρικά και στα πολωνικά. και πάλι σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται η εναρκτήρια συνεδρίαση της ε, σημερινής συνεδρίασης. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, καλώ τους ομιλητές ε, στο τμήμα ε, περί θεσμικής ισορροπίας και διοργανικής συνεργασίας. Θα ήθελα να καλέσω τον καθηγητή Κουάδρος από το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, ο οποίος θα παρουσιάσει τους άλλους ομιλητές. Δεν έχουμε τώρα διάλειμμα για καφέ. Περνάμε κατευθείαν στην, συνεδρία, στην πρώτη συνεδρία της συνδιάσκεψης.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 Κυρίες και κύριοι, με την αδειά σας. C'est Κυρίες και κύριοι, θα κηρύξουμε την έναρξη της πρώτης συνεδρίας της σημερινής συνδιάσκεψης. Θα ήθελα τώρα να κάνω κάποιες πρώτες παρατηρήσεις. Παρακαλώ, θα ξεκινήσουμε, οπότε καθίστε παρακαλώ. Όπως σας είπα, θα ξεκινήσουμε την πρώτη συνεδρία και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτα-πρώτα θέλω να χαιρετήσω τους παρόντες, την κυρία Επίτροπο Βασιλείου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους επιτρόπους, τους ε, διπλωματικούς εκπροσώπους που βρίσκονται εδώ και τους ε, ε, αξιότιμους συναδέλφους μου που ήρθαν από διάφορα μέρη του κόσμου. Επίσης θέλω να σας συγχαρώ για τη διοργάνωση αυτής της συνδιάσκεψης. Δεδομένου ότι έχει ως αντικείμενο το θέμα αυτό στην παρούσα στιγμή με το περιεχόμενο που έχει. Η συνθήκη της Λισαβόνας ουσιαστικά επανειδρύει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την ίδρυση, αν προτιμάτε, μιας νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει μια νέα όθηση στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε, κάποια, σε αυτή τη στιγμή όπου έχει προχωρήσει η παγκοσμιοποίηση και κυρίως σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζει η Ευρώπη από οικονομικές απόψεις, όπως μας εξήγησε ο, Επίτροπο, ο Πρόεδρος Μπαρόζο. Θα ήθελα να επαναλάβω τα συγχαρητήριά μου, τα συγχαρητήρια τα οποία απευθύνω κατά πρώτο λόγο στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσωπική του δέσμευση για την διοργάνωση αυτής της συνδιάσκεψης και θεωρώ σκόπιμο να πω ότι η διοργάνωση μιας τέτοιας συνδιάσκεψης πρέπει να ερμηνευθεί ως αναγνώριση των μεγάλων υπηρεσιών που παρέχει το πρόγραμμα Ζωμονέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τώρα μετά από αυτό θα ήθελα να ευχηθώ, να εκφράσω την ευχή να διατηρήσει την αυτονομία του το πρόγραμμα Ζωμονέ και να κερδίσει περισσότερη ε, ζωτικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Δικυρός που ε, με κάλεσε να προεδρεύσω αυτή τη συνεδρία και θέλω να την ευχαριστήσω για το έργο το οποίο κάνει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Είναι προνόμιο για μένα που προεδρεύω αυτή την στρογγυλή τράπεζα με παρουσία διακεκριμένων προσωπικότητων που συνδέονται εδώ και καιρό με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ε, πω ένα τελευταίο, μια τελευταία λέξη για το περιεχόμενο αυτού του θέματος αυτής της συνεδρίας. Σε όλες τις αναθεωρήσεις των συνθήκων, η θεσμική ε, μεταρρύθμιση και η θεσμική ισορροπία ή πολλές φορές ο απολογισμός μεταξύ των οργάνων ήταν ένα θέμα που ε, έτυχε δύσκολης διαπραγμάτευσης. Δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι κατά την εκπόνηση της ε, συνταγματική συνόδου και πιο μετά της ε, μεταρρυθμιστικής συνόδου οι διαπραγματεύσεις έγιναν πιο δύσκολες με δεδομένες τις καταστάσεις του 2004-2007 που άλλαξαν τις ισορροπίες μεταξύ των μεγάλων, μεσαίων και μικρών κρατών. Πιστεύω ότι αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης ε, σήμερα και της θεματολογίας μας και θα το δούμε στην πράξη. Η δυσκολία προκύπτει στο αντικείμενο αυτό ε, και αφορά ε, όχι μόνο βέβαια τη σύνθεση της Κομισιόν, κυρίως όμως αυτή την τροποποίηση του συστήματος στάθμισης ψήφου στο Συμβούλιο, τον τρόπο υπολογισμού της ε, ειδική πλειοψηφίας και κατ' επέκταση και της ε, δεσμευτικής μειοψηφίας και βεβαίως για τα νομικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής υπόθεσης. Βεβαίως, ε, δεν θα επεκταθώ σε αυτό το θέμα, ούτε θα καθυστερήσω, ε, δεν θα σας ε, δεν θα παρατείνω κατά κάποιο τρόπο την αναμονή σας για να ακούσετε τους επόμενους ομιλητές. Ήδη γνωρίζετε τους επόμενους ομιλητές. Για τις ε, πολιτικές προοπτικές ε, θα ακούσουμε τον κύριο Μάρου Σεφκοβιτς που είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ασχολείται με θέματα διοίκησης και οργανικά θέματα και τον κύριο Κόρμπατς που είναι αντιπρόσωπος μέλος του γραφείου της του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα, από ακαδημαϊκής απόψεως θα ακούσουμε τον κύριο Μόραρ του Τμήματος ε, Διοικητικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο Κολέγιο της Ευρώπης ε, και κάτοχος έδρας ε, Jean Monnet ε, στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, την κυρία Σερένα Ρώση, έδρα Ζωμονέ και ε, Διευθύντρια του Κέντρου Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και τέλος τον κύριο Φερδινάντο Ρικάρντι, ε, εκδότη του περιοδικού Agence Europe. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Σεύκοβιτς. Ευχαριστώ καθηγητά γιατί προφέρατε άψογα το όνομά μου. Μπράβο σας και ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την αγαπητή συνάδελφο Αντρούλα για τη διοργάνωση αυτής της διάσκεψης. Το εκτιμώ ιδιαίτερος γιατί έχουμε πολλούς ευρωβουλευτές, πολλούς πρέσβεις και πολλοί καθηγητές δέχτηκαν την πρόσκλασή μας για να, για να κάνουμε από κοινού αυτή τη συζήτηση που αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νέο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Ξέρω ότι όλα αυτά τα έχετε ξανακούσει, αλλά πολύ εκτιμώ το έργο των καθηγητών Monnet. Σε ολόκληρο τον κόσμο, με στόχο τη διάδοση ε, της ευρωπαϊκής ιδέας. Και κάνετε ένα έργο διαπαιδαγώγησης, ε, ποια ωφέλη αποφέρει η Ευρώπη για τον πολίτη και θα έλεγα και για τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. γιατί είναι πολύ λεπτή στιγμή και πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Οι διαθεσμικές ισορροπίες, η διαθεσμική συνεργασία σε αυτή τη φάση κατόπιν της Λισαβόνας. Όταν μονατέθηκε το χαρτοφύλλο και του αντιπροέδρου για τις διαθεσμικές σχέσεις, <laughs> γνώριζα ότι θα ήταν μεγάλη πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή, διότι έχω την ευκαιρία από πολύ κοντά να παρακολουθώ τις διαθεσμικές ε, σχέσεις και τη διαθεσμική συνεργασία και τη διοργανική συνεργασία. Και βλέπω τη νέα χαρτογράφηση της Ευρώπης μετά τη Λισαβόνα. Να ξεκινήσουμε από το θεσμικό όργανο που σήμερα μας φιλοξενεί, να πάρουμε πρώτα απ' όλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σαφώς ενισχύθηκαν. Η συναπόφαση είναι πλέον η σύνηθις νομοθετική διαδικασία και πέραν του 90% των νομοθετικών πράξεων εγκρίνονται από κοινού ε, από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Οπότε η δυναμική είναι τελείως καινούρια σε επίπεδο νομοθετικό, σε επίπεδο έγκρισης αποφάσεων στις Βρυξέλλες. Αυτό ισχύει και για τομείς όπου είναι σαφέ, σαφές ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας από πλευράς όλων των θεσμικών οργάνων. Περνάμε στους νέους τομείς δηλαδή της συναπόφασης. Ας πούμε, γεωργία, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις και κάτι ακόμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα δικαιούται άμεσα να ενημερώνεται για τις διεθνείς συμφωνίες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμφωνιών προς έγκριση απαιτούν και τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα και πάλι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύθηκε σε όλους αυτούς τους τομείς. Το Ευρωκοινοβούλιο απέδειξε σαφώς και με συμφωλικό τρόπο αναφέρομαι στην απόφαση περί SWIFT, ότι είναι έτοιμο να αξιοποιήσει πλήρως ε, τις νέες του εξουσίες και να παίξει το ρόλο του συνομοθέτη πολύ σοβαρά. Διότι τώρα το Κοινοβούλιο δουλεύει πραγματικά επί ίσης όρης, μαζί με το Συμβούλιο όταν μιλάμε για θέματα νομοθετικά και δημοσιονομικά. Εγώ ήμουν ο διαπραγματευτής εξ ονόματος της Κομισιόν για την επίτευξη της νέας διοργανικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Ποιο είναι ο μοναδικός μου στόχος της ε, διαπραγματεύσεις αυτές. Το Ευρωκοινοβούλιο να φέρει πέρα στην αποστολή του όπως προβλέπεται από τη συνθήκη ούτω ώστε να ενισχυθεί η κοινοτική μέθοδος και οι διοργανικές ισορροπίες. Να περάσουμε στο συνομοθέτη, στο Συμβούλιο έχω την τιμή να παρακολουθώ τις εργασίες του Συμβουλίου γιατί εκπροσώ την Κομισιόν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που όπως γνωρίζετε φέρει την ευθύνη για οριζόντια θέματα αλλά επίσης και για τις προπαρασκευαστικές εργασίες των Ευρωπαϊκών Συνόδων Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχουμε, γίνονται κάμποσες τέτοιες σύνοδοι κορυφής πρόσφατα, θα το έχετε προσέξει. Εδώ και αν ε, βλέπουμε τη νέα η ειδική πλειοψηφία πλέον απολυτελεί τη σύνηθη διαδικασία. Κάνω τη σύγκριση με τον καιρό που ήμουν εγώ μόνιμος αντιπρόσωπος της Σλοβακίας στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσωπών για μια πενταετία, τώρα η δυναμική έχει αλλάξει εντελώς. Τα κράτη-μέλη τώρα δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από την αρνήση κυρία. Όχι, οφείλουν να παρουσιάσουν σαφή επιχειρηματολογία και να είναι πιστική επιχειρηματολογία. Όταν το Συμβούλιο θα εξοικειωθεί πλήρως με, με το νέο αυτό πλαίσιο, πιστεύω ότι θα είναι ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διαδικασία λήψη αποφάσεων και στο Συμβούλιο τι απαιτείται ένθεν και ένθεν σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου και σε επίπεδο Συμβουλίου. Βαθμιαία θα πρέπει να προχωρήσουν σε προσαρμογές. ούτω ώστε οι συνομοθέτες να εφαρμόζουν σωστά τις νέες διαδικασίες. Ας πούμε, νέος μηχανισμός συντονισμού με στόχο την επίτευξη των συμβιβαστικών λύσεων Όλοι αυτοί οι συντοριστικοί μηχανισμοί είναι κέρια σημασίας για το μέλλον. Μας αναμένουν πολύ λεπτές προκλήσεις, άρα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η νέα κατάσταση με τα νέα δεδομένα, ιδίως σε θέματα προπολογισμού, ιδίως σε θέματα δημοσιονομικά. Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω στους νέους παίκτες σε αυτό το διαθεσμικό παιχνίδι των Βρεξελών να ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χαίρομαι διότι κύριε Κορμπέτ θα πάρετε το λόγο ευθύ αμέσω μετά από μένα. Θα με διορθώσετε αν κάνω λάθο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για πρώτη φορά αποτελεί επισήμω θεσμικό όργανο. Ε, έχει μόνιμο πρόεδρο και δικό του προπολογισμό. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ιδιαίτερα βαρυφορτωμένη ημερήσια διάταξη. αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μόνο μάλιστα, χωρίς ε, υπουργούς, με θέματα της καυτής επικαιρότητα. Δίνει νέα όθηση και ενισχύει περαιτέρω το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το γεγονό αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έπαιξε και θα παίξει και μελλοντικά κέριο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, το έργο αυτό θα πρέπει να σέβεται το κοινοτικό πνεύμα που είναι τόσο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι για μας δεν είναι σημαντικό μόνο ποιες αποφάσεις λαμβάνονται αλλά και πώς λαμβάνονται. Αυτό θα, το θα πρέπει να το έχουμε όλοι μας κατά νου. Περνάμε σε άλλο νέο παράγοντα που πιστεύω ότι όλο και περισσότερο ε, θα καταστεί σημαντικός για τη λήψη αποφάσεων στις Βρυξέλλες εμπλοκή των εθνικών βουλών στην όλη διαδικασία. Από την 1η Δεκεμβρίου, όπως γνωρίζετε, χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας, η Κομισιόν εισήγαγε κάποιες διατάξεις για ένα μηχανισμό ελέγχου της επικουρικότητας που τον ασκούν οι εθνικές βουλές. Τώρα οι εθνικές βουλές δικαιούνται να ελέγξουν κάθε νομοθετική πρόταση της Κομισιόν Δηλαδή, κατά πόσο σέβεται τους κανόνες της επικουρικότητας. Να βεβαιωθούν ότι η Κομισιόν προτείνει το ορθό επίπεδο για τη λήψη αποφάσεων. Το ευρωπαϊκό ή πιστεύουν οι εθνικές βουλές ότι θα ήταν προτιμότερος ο χειρισμός σε εθνικό επίπεδο. Άρα τα ευρωπαϊκά ζητήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έτσι θα έχουμε και καλύτερη ανάδραση από τις πρωτεύουσες προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πώς βλέπουν το έργο μας, πώς βλέπουν τις νομοθετικές μας προτάσεις. Άρα θα ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον διότι δεν θα γίνονται συζητήσεις μόνο σε υπουργικό επίπεδο. Άρα οι υπουργοί θα λαμβάνουν καλύτερες συστάσεις από τις εθνικές τους βουλές. Όπως γνωρίζετε, οι εθνικές βουλές ήδη συμμετέχουν σε εντατικές ανταλλαγές ε, με την Κομισιόν. Αυτό γίνεται ήδη ο πρόεδρος Μπαρόσο και η προκάτοχός μου κυρία Βάλστρομ ανίσχυσαν τον πολιτικό διάλογο, ανέκαθεν ενημερώναμε τις εθνικές βουλές. Και βεβαίως εμείς λαμβάναμε τη γνώμη. Λαμβάνουμε τη γνώμη των εθνικών βουλών. Αλλά τότε δεν υπήρχε βεβαίως ε, νομοθετικός αντίκτυπος. Μπορώ να σας πω ότι Πέρυσι είχαμε 250 τέτοιε νομοδοτήσει από τι Εθνικέ Βουλέ, ενώ προηγουμένω είχαμε μόνο μερικέ δεκάδε. Οπότε προφανώ και δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον οι Εθνικέ Βουλέ για μεγαλύτερη εμπλοκή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αυτό το χαιρετίζω. Το θεωρώ ως πολύ θετική τάση. Από τη στιγμή που εισήγαμε αυτόν τον μηχανισμό ελέγχου της επικουρικότητας, και από τη στιγμή που παρουσιάσαμε τι πρώτε προτάσει κανονισμού ε, στου συνομοθέτες, μέχρι στιγμή φέτο λάβαμε τρει αρνητικές ε, γνωμοδοτήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήδη με τη νέα αυτή διαδικασία ε, μηχανισμού εποπτείας της επικουρικότητα και έξι θετικέ. Είμαι βέβαιος ότι θα αυξάνονται συνεχώς τα νούμερα Είχα κάποιες επαφές ε, στη Στοκχόλμη με τους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σαφές ότι τώρα οι εθνικές βουλές δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, ιδίως σε νομοθετικό επίπεδο. Άρα τώρα παίζουν ε, νέο ρόλο, ενισχυμένο ρόλο και οι εθνικές βουλές. Βεβαίω έχουμε και την Επιτροπή των Περιφερειών επιστρέφω στι Βρυξέλλε, με ενισχυμένε επίση εξουσίε, χάρη στη συνθήκη τη Λισαβόνα, και δικαιούνται να προσφύγουν ενώπιον του ΔΕΚ σε θέματα όπου απαιτείται η διαβούλευση και η επικουρικότητα είναι ένα εξ αυτών. Να περάσω σε ένα εντελώ καινούριο στοιχείο, νέο στρώμα στο δημοκρατικό μας οικοδόμημα στις Βρυξέλλες μέχρι στιγμής μέλησα για την προσωπευτική δημοκρατία, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις Εθνικές Βουλές. Τώρα χάρη στη συνθήκη τη Λισαβόνα έχουμε ένα νέο στρώμα συμμετοχική δημοκρατίας που είναι οι πολίτε, που είναι η κοινωνία των πολιτών. Είχα την τιμή να παρουσιάσω πρώτα στην Κομισιόν, μετά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά στο Συμβούλιο προτάσεις για την πρωτοβουλία των πολιτών ένα εκατομμύριο πολίτες θα δίνανται να καθορίσουν κάποιο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα είναι μελλοντικά πώς θα αξιοποιηθεί αυτό το μέσο. Είναι περίπλοκο για τον κάθε πολίτη ή όχι. Να σας πω πώς το βλέπω. Ε, υπήρξε, υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον από όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα θα υπάρχει αυτή η επιγραμμική δυνατότητα συλλογής υπογραφών. Ακούω να κυκλοφορούν διάφορα σχέδια, οπότε πιστεύω ότι θα χρησιμοποιηθεί ευρέως μελλοντικά αυτό το μέσο. Οπότε θα υπάρχει μεγάλη πολιτική κινητοποίηση για προώθηση κάποιων θεμάτων στις Βρυξέλλες. Η κοινωνία των πολιτών δίνει μάχη για να, κάνει ακουστή τη φωνή της με βάση το άρθρο 11 το περίφημο της συνθήκης της Λισαβόνας για μίλα για μεγαλύτερη συμμετοχή της στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και χρησιμοποιούμε κάθε δυνατή δίωδο μέσα των οικονομικών επιτροπών για την ενίσχυση αυτού του διαλόγου μας με την κοινωνία των πολιτών και φαντάζομαι ότι μελλοντικά θα έχουμε και περαιτέρω ενίσχυση. Άλλος πολύ σημαντικός νέος παράγοντος είναι η υπηρεσία των εξωτερικών σχέσεων, αλλά αυτό προβλέπεται σε άλλη σύνοδο Απλά σας λέω ότι με την Κάθι Ένστον έχουμε εξαιρετική συνεργασία, πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και με το Συμβούλιο και με το Ευρωκοινοβούλιο και ελπίζω ότι θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Διπλωματική Υπηρεσία άμεσα, διότι το χρειαζόμαστε για να μιλάμε με μία φωνή, για, για στόχους ενισχυμένης συνοχής και για την προώθηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων στο εξωτερικό. Δουλεύουμε σκληρά προς την επίδευξη αυτού του στόχου και ελπίζω να έχουμε θετική έκβαση. Ιδού το όλο πλαίσιο της ε, διοργανικής διαθεσμικής ζωής της Βρυξέλλες, αλλά άφησε κατά μέρο την Κομισιόν. Τι μένει για την Κομισιόν στην νέα αυτή χαρτογράφηση. Έχουμε περισσότερους παίκτες στο διαθεσμικό παιχνίδι, κάποιοι ενισχύουν το ρόλο τους, η Κομισιόν όμως θα πρέπει να παραμείνει ο θεματοφύλακας ε, της Ένωσης, ε, ο εκπρόσωπος της κοινωνικής μεθόδου, ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας θα αξιοποιηθεί για να εξέρθει τη ύφεση η Ένωση, να ξαραμπεί στην οδό της επιμερίας και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, κάθε τρόπο στο τη οικονομική και επέκταση των πλεονεκτομάτων της ενιαίας αγοράς πανευρωπαϊκά. Πώς, πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις εφαρμόζοντας σωστά τη στρατηγία ε 2020 και ενισχύοντας το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Διότι πάνε χέρι-χέρι και θα πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος και στα δύο μέτωπα. Η Κομισιόν βεβαίω λειτουργεί σε πιο απαιτητικό περιβάλλον με περισσότερου και ενισχυμένου παίκτε. Άρα, η Κομισιόν σοφά θα πρέπει να αξιοποιήσει τις εξουσίες της, ας πούμε, την νομοθετική πρωτοβουλία. Έχει μία διαφυσβήτητη πραγματογνωμοσύνη. Είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο που μπορεί να σας δώσει σφαιρική άποψη της κατάστασης και μάλιστα πανευρωπαϊκά για συγκεκριμένα θέματα. Κανένα άλλο θεσμικό όργανο δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Ε, όλοι εκτιμούν το έργο της Κομισιόν. Έχουμε τεχνική πραγματογνωμοσύνη και θα πρέπει να την εξοπλίσουμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η Κομισιόν ε, και αν εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα άρα θα πρέπει ε, περαιτέρω να διαφυλάξει το σεβασμό του κοινοτικού κεκτημένου Κομισιόν. Εν κατακλείδη, να τονίσω ότι παρά την ποικιλομορφία στο νέο θεσμικό πλαίσιο, αυτό που προέχει για όλους τους φορείς είναι να αντιληφθούν ότι έχουμε ένα στοιχείο από κοινού. Θέλουμε πιο δημοκρατική, πιο ανταγωνιστική, καλύτερη Ευρώπη που να τη σέβονται όλοι στο διεθνές προσκήνιο. Καμιά φορά είναι καθόδης βέβαια οι διαθεσμικές μας συζητήσεις. Είναι όμως σαφές ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά έργανα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν ε, είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι στο DNA βεβαίω όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και αυτή η τάση ελπίζω να επιβεβαιωθεί μελλοντικά. Εν κατακλείδη να αναφέρω το εξή. Είμαι βέβαιος ότι το νέο αυτό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η συνθήκη της Λισαβόνας θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τις νέες εξουσίες όλων των θεσμικών οργάνων προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος των πολιτών της. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup, Monsieur Sefcovic. J'espère que c'est prononcé aussi bien cette fois. Nous, je donne la parole maintenant à Monsieur. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Κόρμπετ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε να είμαι εδώ σήμερα παρόν. Ο κύριος Δεκουάδρας στα εισαγωγικά του σχόλια αναφέρθηκε στη στην συνθήκη της Λισαβόνας ε, ως μια επανίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια νέα ένωση που αντικαθιστά την παλαιά. Αυτό είναι νομικός ορθό πολιτικός όμως, ε, εγώ θα το έβλεπα ως εξέλιξη. Δηλαδή ένα ακόμη βήμα σε μια σειρά βημάτων που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες με συνεχόμενες μεταρρυθμίσεις και στην, ε, στις διοργανικές ε, δομές μέσω της του Μάστριχ, της ενίας πράξης, την συνθήκη της Νίκης, της, τώρα της Λισαβόνας. Μιλώ για μια εξέλιξη βήμα-βήμα, ειδικά σε διαφορά τα θεσμικά, γιατί η συνθήκη τη Λισαβόνα δεν έχει κάνει καμιά ιδιαίτερη αλλαγή σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρμοδιότητες δεν έχουν διευρυνθεί τόσο πολύ. Αυτό που έχει κάνει όμως είναι ο τρόπος με τον οποίο ασκούμε τι αρμοδιότητε που, τις αρμοδιότητες που μας δίνονται μέσω των θεσμικών δομών και των διαφόρων αξιών που έχει το κάθε θεσμικό όργανο. Αυτές είναι οι αλλαγέ που μεταρρύθμισε η συνθήκη τη Λισαβόνα, με έναν διτό στόχο, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη δημοκρατία, περισσότερη δημοκρατία. Ίσως ένα παράδειγμα να σας πω, γιατί μιλώ για βήμα-βήμα, για την εξέλιξη βήμα προς βήμα. Ε, αν δούμε έτσι πιο μακροπρόθεσμα τα πράγματα, θα δούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν πρόκειται για νομοθεσία είχε ρόλο κυρίως συμβουλευτικό μέχρι την συνθήκη του Μάστριχτ η οποία εισήγαγε την ε, διαδικασία της ε, συναπόφασης για πολύ λίγα πάλι άρθρα και ήταν και μια πολύ περιορισμένη αυστηρή διαδικασία τότε. Η διαδικασία αυτή άλλαξε προ όφελο του Κοινοβουλίου με τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογή του, το οποίο διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο με την Νίκαια και τώρα με την Λισαβόνα έχουμε εξουσία ε, ως Κοινοβούλιο σχεδόν σε όλους τους τομείς της νομοθεσίας ε, γιατί μιλούμε για συναπόφαση με το Συμβούλιο. Έγινε λοιπόν βήμα-βήμα όλο αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τις εξουσίες ε, του Κοινοβουλίου για την ε, επικύρωση διεθνών συμφωνιών. Ξεκίνησα με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις συνθήκες προσχώρησης. Έγιναν αλλαγές στις ευρωπαϊκές συνθήκες και αυτό διευρύνθηκε. Πάλι βήμα-βήμα. Και τώρα οποιαδήποτε συνθήκη, οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία συμφωνία που είναι σημαντική χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να επικυρωθεί. Και αυτό επίσης το βλέπουμε και στην Κομισιόν και στην λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν οριζόταν από τις εθνικές κυβερνήσεις για μια τετραετία. Μετά, βήμα-βήμα, και με το Μάστριχ, το Άμστερνταμ, τη Λισαβόνα. Άλλαξε αυτό. Τώρα έχουμε την Κομισιόν που ορίζεται για πέντε χρόνια, δηλαδή συμπίπτει με την θητεία του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβουλίο έχει το, την εξουσία να εγκρίνει την, το διορισμό του, του, της Κομισιόν με την ψήφο εμπιστοσύνη. και με την αλλαγή με τη συνθήκη έπρεπε να, εγκρίνει την επιλογή του Προέδρου και τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας το Κοινοβούλιο, όπως λέει, εκλέγει τον Πρόεδρο της Κομισιόν. Έναν Πρόεδρο ο οποίος μέσω διαφόρων αλλαγών των συνθήκων τώρα έχει το δικαίωμα να δίνει τα χαρταφυλάκια, να κάνει ένα σχηματισμό αν θέλει και να απολύσει ένα μέλος της Επιτροπής. Αυτές λοιπόν ήταν βασικές αλλαγές που έκανε η Λισαβόνα, που έφερε η Λισαβόνα. Προς το παρόν, θα δούμε πόσο θα κρατήσει μέχρι να γίνει η επόμενη αναθεώρηση. Τώρα, αυτό στο οποίο θα ήθελα εγώ να επικεντρωθώ είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κύριος Σεύκοβιτς, αυτό είναι πλέον ένα θεσμικό όργανο δυνάμει τη συνθήκη. Και αυτό έχει τι συνέπειε του. Πρέπει να εγκρίνει τα πρακτικά των συνεδριασεών του. Έχει προπολογισμό, έχει κανόνε εσωτερικού, διαδικαστικού. Μπορείτε να δείτε λοιπόν πώ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ε, έχει ε, ιστοσελίδα, όπως είπε ο κύριος Σεφκοβιτς, δεν ε, παρίστανται οι Υπουργοί Εξωτερικών, μόνο η Καθιάστον βρίσκεται εκεί, η εκπρόσωπο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική κάτι που, είναι, που το καθιστά πιο συγκεκριμένο, πιο δεμένο, λίγο πιο κολυγιακό ε, όργανο. Η πιο μεγάλη όμως αλλαγή έγινε στον πρόεδρο. Πάντα είχαμε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τι άλλαξε. Τρεις μικρές αλλαγές, αλλά συνολικά δημιουργούν μια νέα, ένα νέο σημείο εφετερίας. Η πρώτη αλλαγή ήταν αυτή της συνέχειας. Στο παρελθόν η Προεδρία άλλαζε κάθε δεύτερη ή τρίτη, ε, κάθε έξι μήνες. Με θητεία δυόμιση ετών για κάθε πενταετία ώστε να, γίνεται, να είναι δυνατή η τριτη καθε εξι μηνες με θητεια σχέσεων, να ξέρει κανείς πότε είναι σωστό να μπει κάτι στην ημερήσια διάταξη, όχι να βιάζεται επειδή θα δλήξει η θητεία του, αλλά με βάση την σωστή χρονική στιγμή. Μεγαλύτερη λοιπόν ε, συνέχεια σε ό,τι αφορά τι εξωτερικέ σχέσει μα με τι τρίτες χώρες ή χώρε, η ομάδε χωρων Κορυφής Ευρώπης Λατινικής ευρωπης λατινικη Αμερική. Μερικέ φορέ είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν διαφορετικό πρωθυπουργό κάθε φορά. Τώρα υπάρχει συνέχεια σε αυτό. Δεύτερη αλλαγή. Οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων στο Συμβούλιο μπορούν να επιλέξουν ποιον θέλουν να προεδρεύει των συνεδριάσεων τους και να τους εκπροσωπεί. Όλο λοιπόν αυτό το σύστημα της αυτόματης ε, ε, εναλλαγής δημιουργούσε μία ε, ατμόσφαιρα λοιπούς εμπιστοσύνης γιατί πολλέ φορέ ε, στα πλαίσια τη θητεία του ένα πρόεδρο είχε να αντιμετωπίσει εσωτερικέ ε, εκλογέ στη χώρα του και δεν ήξερα καν αν θα επανεκλεγεί. Τώρα μπορούμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις, ε, όλα αυτά τα προσκόμματα, επιλέγοντα όμω κάποιον. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και ένα βαθμό εμπιστοσύνη. Να υπάρχει δηλαδή μια πολιτική εντολή για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίο επιλέγεται. Η τρίτη αλλαγή είναι ότι αυτό το άτομο έχει πλήρη απασχόληση. Οι παλαιότεροι προκάτοχοι της θέσης αυτής ε, είχανε, έπρεπε να διοικήσουν και τη δική τους κυβέρνηση που προφανώς 80%-90% του χρόνου τους ήταν αφιερωμένο σε αυτό. Τώρα, έχοντας κάποιον με πλήρες ωράριο ως πλήρες ως πρόεδρο, είναι καλύτερο να, γιατί μπορούμε να έχουμε καλύτερη σχέση με κάθε έναν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που αποτελούν το Συμβούλιο. Μπορούν να μιλούν, μπορούν να ε, ταξιδεύουν για να συναντηθούν. Και αυτό λοιπόν είναι μια σημαντική αλλαγή. Αυτές οι τρεις αλλαγές συνολικά θα πρέπει να κάνουν ε, καλύτερη την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και Βέβαια, εντάξει, και αυτό θέτει διάφορα ερωτήματα. Μιλούμε δηλαδή τώρα για ενίσχυση της διακυβερνητικής πλευράς α, τον, του Συμβουλίου έναντι της πιο κοινοτικής πλευράς. Καταρχήν, οι διακυβερνητικέ πτυχές της Ένωσης είναι μια πραγματικότητα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δουλεύει καλά στο σύνολό της και αυτή η πτυχή πρέπει να λειτουργεί καλά, πρέπει να λειτουργεί καλύτερα. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το βήμα στο οποίο συγκερνώνται όλες αυτές οι ε, απόψεις. Είναι το μέρος όπου μπορεί κανείς να συντονίσει και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις πολιτικές. έχουμε, έχοντας έναν πρόεδρο ο οποίος δεν προσπαθεί να υπονομεύσει την κοινοτική πτυχή. Ίσα ίσα ο πρόεδρος Φαν Ρομπάι θέλει να την ενισχύσει την πτυχή αυτή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν δεν προσπαθεί να ηγηθεί στα συντρίμια, στα ερήπια των υπολοίπων οργάνων. Βεβαίω όταν συνετάχθη η συνθήκη υπήρχαν ε, αρκετά προβλήματα, γι' αυτό και δεν υπήρχε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια για το τμήμα αυτό. Υπήρχαν κάποιοι που είδανε, θεώρησαν ότι θα υπάρξει ένας πρόεδρος όπως υπάρχει στην ε, Γαλλία και ότι η ε, και ο πρόεδρος της Κομισιόν θα είναι σαν ε, ένας πρωθυπουργό της Γαλλίας που έχει να κάνει, ασχολείται με εσωτερικά θέματα και τα υπόλοιπα τα σημαντικά τα αφήνει για τον πρόεδρο. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι ήταν τελείως αντίθετο, ότι ήταν πολύ ρεαλιστικό να έχουμε μια συνέχεια στην Προεδρία. Ο πρόεδρος Φαν Ρομπόη ήταν πολύ τα αυτό. Ούτε πρόεδρος στα πλαίσια της γαλλικής δημοκρατίας είναι, ούτε πρόεδρος πρωθυπουργός. Ένας α, δημοσιογράφος πρόσφατα τον κατηγόρησε ότι είναι ένας απλός παρατηρητής και ένας άλλος τον κατηγόρησε ότι έκανε πραξικόπημα. Ένας, ο ίδιος είπε ότι ούτε παρατηρητής είμαι, ούτε δικτάτορας. Είμαι αυτός που διευκολύνει. Και έχοντας υπόψη ότι προεδρεύει του μοναδικού θεσμικού οργάνου που πρέπει να λειτουργεί με ομοφωνία, 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, 27 άτομα που στα, εθνικό τους, ε, στα εθνικά πλαίσια περνάνε την άποψή τους και υπερισχύει η δική τους άποψη, ε, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα άνθρωπο που να μπορεί να δημιουργήσει αυτή την ε, ομοφωνία, να μπορεί να δημιουργήσει γέφυρε μεταξύ ανθρώπων που ξεκινούν από τελείως διαφορετικές οπτικές γωνίες. Βεβαίως πολλά εξαρτώνται και από τι σχέσει με, με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Ο πρόεδρο πρέπει να δημιουργήσει αυτέ τι ε, σχέσει. είναι σε επαφή με πρόεδρου άλλων θεσμικών οργάνων συχνά. Ξέρω ότι τελειώνει και ο χρόνο μου, αλλά ίσω καλό θα ήταν να τα περάσω έτσι, να τα διατρέξω λίγο γρήγορα τα σημεία αυτά, Πρόεδρε. Οι σχέσει λοιπόν με την Βαρόνη Άστον δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Επιπέδου είναι ο διαχωρισμός ε, μεταξύ δηλαδή Προέδρου ή ε, Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών του. Αν η διάσκεψη είναι σε υπουργικό επίπεδο, ε, να προεδρεύει η κυρία Άστον. Αν ε, είναι σε ανώτερο επίπεδο, τότε προεδρεύει ο Πρόεδρος Φανρομπόη. Οι σχέσεις τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπόφευκτα είναι λίγο πιο ευαίσθητες. Η κοινή γνώμη, τρίτες χώρες δεν κατανοούν άμεσα τη διαφορά μεταξύ του Πρόεδρου της Κομισιόν και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οι δύο στις Βρυξέλλες βρίσκονται. Εξωτερική εκπροσώπηση και οι δύο εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και οι γραμμές εδώ, οι διαχωριστικές δεν είναι απόλυτα σαφείς πάντα. Στο επίπεδο τη Κάθιαρστον έχουμε ενώσει την εκπροσώπησή μα και έχουμε ε, τις, ε, τις θέσεις που είχε ο κύριος Σολάνα και ο κύριος Πάτον και έχουμε φτιάξει την κυρία Πατάνα, δηλαδή την κυρία Άστον που εκπροσωπεί την ε, Ένωση. Αλλά έχουμε τονίσει τη διαφορά. Και δεν θα με εκπλήξει αν σε λίγα χρόνια έχουμε μια συζήτηση που θα μιλά πάλι για επανένωση θέσεων. Εν τω μεταξύ όμω αυτό το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει. Οι δύο πρόεδροι γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρέπει να βοηθήσουν, πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα, πρέπει να αποφύγουν τους, ε, τις μάχες μεταξύ τους. Γι' αυτό συναντώνται κάθε Δευτέρα για πρωινό. Ενήλικες είναι, ξέρουν πώς δουλεύει το σύστημα, ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να λειτουργήσει. Σχέσεις τώρα με το Κοινοβούλιο. Η το μόνο καθήκον του Προέδρου δυνάμει της συνθήκης είναι να δίνει αναφορά στο Κοινοβούλιο μετά από κάθε ε, συμβούλιο για 5-6 φορές το χρόνο ας πούμε. Αυτά. Ε, ο πρόεδρος ε, ήθελε να το συμπληρώσει αυτό και το έκανε. Έχει συναντήσει τους πρόεδρους των πολιτικών ομάδων, των επιτροπών. Το κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα δέχτηκε την πρόταση του Προέδρου Φανρομπόη να ενημερώσει τους αρχηγού όλων των πολιτικών ομάδων αμέσω μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μάλιστα με το ίδιο απόγευμα, μόλις τελειώσει το Συμβούλιο, να τους δώσει ζεστέ πληροφορίες για το τι έγινε. Θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχει σχέση με το Κοινοβούλιο, αλλά δεν θέλει να υποκαταστήσει ε, το, τον πρόεδρο της Κομισιόν. Ο πρόεδρος της Κομισιόν έχει πιο στενή σχέση με το Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος της Κομισιόν είναι υπόλογος στην, ε, στο Κοινοβούλιο και μπορεί να απο, αποπεμφθεί και από το Κοινοβούλιο. Υποβάλλει το σχέδιο προπολογισμού στο Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρο ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν κάνει τίποτα. Είναι λοιπόν άλλη η σχέση του με το Κοινοβούλιο. Και τέλο, ποια είναι η σχέση με την ε, εκπεριτροπής προεδρία. Η εκπεριτροπής προεδρία θα είναι άλλη ιστορία. Η Ισπανική Προεδρία σε πολλούς, με κατά κάποιο τρόπο ήταν η τελευταία του συστήματος αυτού. Από εδώ και στο εξή, η εκπεριτροπή Προεδρία δεν θα, ο πρόεδρος μάλλον της ο Πρωθυπουργός δεν θα ε, προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ούτε ο Υπουργός Εξωτερικών θα προεδρεύει του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. τα θέματα τώρα της ε, προσώπησης στο εξωτερικό ε, των, ε, της εξωτερικής πολιτικής τα έχει αναλάβει η κυρία Άστον. Ούτε οι πρεσβείες θα έχουν να, να συντονίσουν τις πρεσβείες της υπόλοιπες χώρες. Η Εκπαιδευτική λοιπόν Προεδρία απλώς θα είναι η Προεδρία των τομεακών ε, συμβουλίων ε, γεωργίας, ε, μεταφορών, περιβάλλοντος. Γιατί εκεί υπάρχει συνομοθεσία με το κοινοβούλιο. Δεν θα έχουν λοιπόν το ρόλο που είχαν πριν. Βέβαια, εντάξει, και πριν είχαν πάλι την επιτροπή, την προεδρία, συγγνώμη, ενό συγκεκριμένου τομέα για έξι μήνε με συγκεκριμένη μερίσια διάταξη και χωρί καμία άλλη εξουσία. Απλώ προέδρευαν μια συνεδρία, μια υπουργική ε, διάσκεψη. Τώρα θα είναι ακόμη λιγότερο σημαντικό ο ρόλο του. Και αυτό δεν το έχουν συνηθίσει πολύ. Και κάποιες κυβερνήσεις ε, έχουν ξεχάσει. Έχουν ξεχάσει τι υπήρχε στην συνθήκη που υπέγραψαν. σω το υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση από αυτέ. Αλλά πολλοί θέλουν ακόμη να έχουν έτσι πολύ υψηλό ρόλο και ψάχνουν να βρούνε κάτι για να παραμείνει το κύρος που είχαν από πριν. Είναι λοιπόν αρκετά ευαίσθητα τα πράγματα εδώ για το πώ πρέπει να το διαχειριστούμε. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα. Έτσι θεωρώ εγώ ότι ε, εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εγώ λέω ότι και πάλι ότι είναι εξέλιξη και όχι επανάσταση ε, για την ε, μετέπειτα λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά την δημοκρατική της ευθύνη και την αποτελεσματικότητά της. Ευχαριστώ. Ακούσαμε δύο πολύ ξεκάθαρες και πλούσιες παρουσιάσεις, ακόμη και αν διέφεραν ως προς το περιεχόμενο για τις πολιτικές προοπτικές της θεσμικής ισορροπίας. Τώρα περνάμε στην ακαδημαϊκή προοπτική και θα δώσω το λόγο πρώτα-πρώτα στον κύριο Γιώργο Μονάρ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που είμαι σήμερα εδώ για να σας μιλήσω για το θέμα της θεσμικής ισορροπίας. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεκουέρος ε, για την πρόσκληση, την οποία δέχτηκα με ιδιαίτερη χαρά. Θα χρησιμοποιήσω κάποιες διαφάνειες PowerPoint για την παρουσίασή μου και δεν θα τις ε, κάνω, δεν θα τις χειριστώ εγώ, θα πρέπει να δίνω κάποιο σήμα και ζητώ συγγνώμη για τις ε, όποιες διακοπές. Πρώτη διαφάνεια παρακαλώ. Πρώτα πρώτα πρέπει να σας ξεκαθαρίσω πώς εννοώ εγώ τη χρήση της θεσμικής ισορροπίας. Υπάρχουν δύο όροι. Υπάρχει η θεσμική ισορροπία ως θεσμική ε, αρχή. Τώρα εδώ μιλάμε για την κατανομή των εξουσιών. Ε, αυτή η κατανόηση, αυτή η έννοια έχει αναπτυχθεί από το ΔΕΚ ε, σε αρκετές υποθέσεις. Ξεκίνησε ήδη η περιπόθεση C56 μερώνει και καθόρισε την ε, έννοια αυτή ως στόχο την προστασία των προνομίων όπως αυτά ορίζονται ε, στις συνθήκες. Η διάκριση αυτή ε, της έννοιας χρησιμοποιείται και στη βιβλιογραφία και στις πολιτικές επιστήμες και υπάρχει και η έννοια της θεσμικής ισορροπίας ως η σχέση μεταξύ των φορέων. Υπ' αυτή την έννοια στηρίζεται στις σχετικές εξουσίες των θέσεων εντός των διαφόρων φορέων εντός ενό συγκεκριμένου πλαισίου. Εδώ έχουμε μια δυναμική έννοια, διότι πρόκειται για ε, διασύνδεση εξουσιών μεταξύ των φορέων από τη δεκαετία του 50 και εγώ θα εστιάσω την προσοχή μου στην παρουσίασή μου στη δεύτερη έννοια, ε, δηλαδή των σχέσεων εξουσιών και θα δούμε τι ακριβώς άλλαξε με τις συνθήκες της Λισαβόνας και ποιες θα είναι και οι πιθανές επιπτώσεις. Η επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Ήδη ε, ο Επίτροπος Εύκοβιτς ε, είπε ότι τα πράγματα άλλαξαν ε, ξεκάθαρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και ο κύριος Κόρμπετ επεσήμανε την αύξηση της εξουσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την ε, αρχή του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, από τη δεκαετία του 70, από τότε που το Κοινοβούλιο έλαβε τις πρώτες δημοσιονομικές εξουσίες, είχαμε ένα διπολικό σύστημα. Δηλαδή, αν δείτε και τα παλιά κείμενα στη βιβλιοθήκη του Κολεγίου της Ευρώπης, γιατί τα κρατάμε τα παλιά βιβλία για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ε, όπου χρησιμοποιούνται ο όρος θεσμική ισορροπία εννοείται κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αργότερα μπήκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ευρωπαϊκό Σύστημα και από το 70 και μετά γίνεται ε, όλο και περισσότερο λόγος για ένα τρίπολικό σύστημα, δηλαδή Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο βέβαια ήταν στην αρχή, στο πάνω μέσα στην κορυφή του ε, τριγώνου αυτού. Το έβαλα εκεί για να απονείμω τιμή, φοροτιμή στους ε, ε, οικοδεσπότες μας σήμερα εδώ. Ε, υπάρχει και ένα υβριδικό τέτραπολικό σύστημα και περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ λοιπόν Έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο όπως σας εξήγησα μπαίνει στο σύστημα από νομικής και συνταγματικής πλευράς ε, ως πλήρες ε, όργανο με τη δυνατότητα να, θεωρεί, να υιοθετήσει νομικά δεσμευτικές αποφάσεις και βεβαίως ε, και το κόστος και για τις δαπάνες υπόκειται σε θεσμικές ε, κατά κάποιο τρόπο ε, υποχρεώσεις για την θεσμοθέτηση της διαφάνειας. Ε, πολλές φορές θα μπορούσε να προσβληθεί και ενώπιον του δικαστηρίου και συνέβη αρκετές φορές αυτό. Και στο κάτω μέρος του τριγώνου, στο κάτω τρίγωνο αυτού τετραπολικού συστήματος μπορείτε να δείτε ένα νέο πολύπλοκο σύστημα που έχουμε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι και ύπατη πρόσωπος. Εδώ έχουμε ένα είδος, και εδώ είναι μεγάλη καινοτομία, ένα είδος υποτρίγωνο των εξουσιών το οποίο προέκυψε και το οποίο περιβάλλει τη νέα θέση και δεν πρόκειται για μια νέα ακριβώς θέση που δημιουργήθηκε, αλλά υπάρχει και μια διοικητική μηχανή που την υποστηρίζει και υποστηρίζει τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη νέα συνθήκη λοιπόν έχουμε λίγο πολύ ρητά σχέσεις καθορισμένες ε, σχέσεις εξουσίας μεταξύ των διαφόρων οργάνων τα οποία βρίσκονται στο διάγραμμα αυτό αλλά ε, η λιγότερο προσδιορισμένη σχέση είναι αυτή μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εδώ δεν έχουμε ιεραρχική σχέση, δεν έχουμε άμεσες μορφές αλληλεπίδρασης και διάδρασης ε, και αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον, ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό το οποίο δεν βρίσκεται συνήθως σε εθνικές θεσμικές διοργανώσεις. Επόμενη διαφάνεια. Η, η θεσμική ισορροπία λοιπόν. Θα διατρέξω εντρά, εντάχει. Μπορούμε να διακρίνουμε έξι διαστάσεις της ισορροπίας αυτής. Πρώτον, συνταγματική θέση, δηλαδή η θεσμική αυτονομία των οργάνων, τις εξουσίες για τις αλλαγές των συνθήκων, τις, τα δημοσιονομικά θέματα και τις ε, βασικές, ε, την, ε, τις βασικούς διορισμούς. Εκκίνηση πολιτικής επίσης, προγραμματισμός και νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τέταρτο στοιχείο είναι η λήψη αποφάσεων δηλαδή πρωτογενείς νομοθετικές και δημοσιονομικές εξουσίες. Μετά έχουμε την εφαρμογή τι εξουσίες δηλαδή έχουν τα όργανα για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται, μεταξύ των οποίων και έλεγχο της εφαρμογής από τα κράτη-μέλη. Μετά έχουμε ε, θεσμική ισχύ, δηλαδή ηγετική σχέση και συνεκτικότητα, διότι βεβαίως όλα αυτά μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην διασύνδεση εξουσιών μεταξύ των οργάνων. Και τέλος, και εδώ θα αποκλίνω από την κοινή έννοια της ισορροπίας. Μιλάμε για την ε, ορατότητα, τη δημόσια ορατότητα. Δηλαδή είναι θεσμοί που είναι περισσότερο ορατοί στις διεθνείς σχέσεις και μπορούν να αυξήσουν την επιρροή τους μέσω της ενισχυμένης ορατότητας και ενώπιον της κοινή γνώμης αλλά και των διαφόρων ε, εταίρων. Τώρα θα δούμε τις διάφορες αυτές διαστάσεις χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Πρώτον, οι αλλαγές ισορροπία σχετικά με τις συνταγματικές θέσεις. Εδώ είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο ε, προκύπτει με πολύ ενισχυμένη θέση από την συνθήκη του Λισαβόνα. Έχει ενισχυμένο ρόλο για την αναθεώρηση ε, των ε, συνθήκων, ρόλο διαπραγματευτικό, ενισχυμένο ρόλο στις διατάξεις ε, περί ευελιξίας για, την, ε, για τα ποινικά θέματα. Έχει αυξημένο ρόλο για την κίνηση της ενισχυμένης συνεργασίας, κάτι που δεν ίσχυε πιο πριν και επίσης και ε, τον διορισμό της Κομισιόν. Εκεί έχει ενισχυθεί η θέση του. Και τέλος επίσης έχει εξίσου με το Συμβούλιο ε, Δημοσιονομικές Εξουσίες. Επομένως η θέση του Κοινοβούλιο ενισχύεται και το Κοινοβούλιο, ε, και εδώ υπάρχει σημαντική αλλαγή. Το Κοινοβούλιο είναι, έχει επηρεαστεί ε, ιδιαίτερα από την αλλαγή αυτή, διότι αυτή η θέση, ο ρόλος ως διαπραγματευτή, διαμεσολαβητή, ε, δημοσιονομική αρχή δίνει στο κοινοβούλιο τη δυνατότητα να επηρεάζει το γίγνεσθε. Ε, το συμπε... Η Κομισιόν βρίσκεται εξασθενημένη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ενισχυμένο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ε, ο ύπατος εκπρόσωπος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, υποστηρίζει την ομοιογένεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά κάποιο τρόπο το Συμβούλιο παίρνει μισή έδρα κατά κάποιο τρόπο στο σώμα των Επιτρόπων. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια σχετική εξασθένηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα από συνταγματικής πλευράς το Συμβούλιο δεν έχει αλλάξει θέση, μόλον ότι γίνεται κάπως πιο είναι κάπως πιο ισχυρό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, έχει ενισχύσει τη θέση του, δεν είναι πλέον μόνο ένας ε, φορέας που συνεδριάζει, αλλά ε, μπορεί να θεσπίσει και νομικά δεσμευτικές αποφάσεις και μπορεί να διορίσει ή να αποπέμψει μέλη της Επιτροπής. τώρα, αλλαγές στην ισορροπία σχετικά με τον τομέα τη εκκίνηση πολιτική. Και εδώ πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κερδίζει περισσότερο από τι αλλαγέ που προέκυψαν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα έμεσα διότι ε, γενικά ενισχύεται η θέση του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχυμένο διάλογο για τις προτα... νομοθετικές προτάσεις και τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση, αλλά τελικά μάλλον το Κοινοβούλιο θα πετύχει κάτι ουσιαστικό. Και ο Πρόεδρος Μπαρόζο ε, ήδη το υποσχέθηκε σε μεγάλο βαθμό. Επομένω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαφώς κερδίζει κάτι από αυτή την πλευρά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως βγαίνει εξασθενημένη, διότι το αποκλειστικό δικαίωμα πρωτοβουλία, και θα δούμε και σε, σε ποιο βαθμό θα γίνει, ε, ουσιαστικά ε, μπορεί η Κομισιόν να υποχρεωθεί από τους πολίτες να υποβάλει μια, να αναλάβει μια πρωτοβουλία που δεν θα είχε αναλάβει διαφορετικά. Οπότε θα πρέπει να πω ότι υπάρχει μια de facto κοινοτικοποίηση του τρίτου πυλώνα, δηλαδή για τα ποινικά θέματα δικαστική συνεργασία. Και εδώ για πρώτη φορά, στην περίπτωση της κοινοτικοποίησης ενός πεδίου πολιτικής, δεν είχαμε πέρασμα σε αποκλειστικό δικαίωμα πρωτοβουλίας της Κομισιόν. Ανταυτού, ένα κράτος μέλος μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα να περιορίσει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αυτό εννοούμε με την ε, κοινοτικοποίηση και κάποιες αποφάσεις μπορούν να ανασχεθούν από το ε, εργαλείο ελέγχου περί ε, επικουρικότητας των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δηλαδή, το, η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντικατασταθεί για το τομέα της ΚΕΠΑ από την δυνατότητα να υποστηριχτούν προτάσεις που υποβάλλει ο ύπατος εκπρόσωπος. Και εδώ βλέπουμε μία μείωση, λοιπόν ελαφρά μείωση του ρόλου πρωτοβουλίας της Κομισιόν. Το Συμβούλιο δεν έχει αλλάξει θέση βασικά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όμως ε, έχει ενισχυμένη θέση διότι αν ε, διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο της συνθήκης, ε, είναι ισχυρότερη η διατύπωση που χρησιμοποιείται για τον στρατηγικό ρόλο προσανατολισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δηλαδή, για παράδειγμα, σχετικά με την ΚΕΠΑ, ε, υπάρχει η έννοια του ορισμού του στρατηγικού συμφέροντος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι το οποίο προσθέθηκε σε κάτι που υπήρχε ήδη στη συνθήκη, στις γενικές κατευθυντήρες γραμμές, στον τομέα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που είναι ε, ε, ήταν ο ευρύτερος τομέας πολιτικής την τελευταία δεκαετία. Στο άρθρο 68 της Συνθήκης της Λισαβόνας μιλά για το ε, ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον καθορισμό του προγράμματος και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο, προβλέπει 82 σελίδες με στόχους και αυτά παραμένουν στο Συμβούλιο. Η επόμενη διαφάνεια, λήψη αποφάσεων. Το Κοινοβούλιο και εδώ κερδίζει στην ισορροπία, έχει επεκταθεί η συναπόφαση, ε, πλήρη συναπόφαση ε, και για τα δημοσιονομικά θέματα που είναι πολύ ισχυρές εξουσίες για τη λήψη αποφάσεων και σαφώς θα κάνουν τη διαφορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγαίνει εξασθενημένη, λόγω της ε, επέκτασης της συναπόφασης. Δηλαδή υπάρχουν 40 περίπου νέοι τομεί όπου θα πρέπει να συνυπολογίσει το Κοινοβούλιο στην ε, νομοθετική διαδικασία και αλλάζει, επηρεάζεται λοιπόν το δικαίωμα πρωτοβουλία της ευρωπαϊκή Επιτροπής σημαντικά. Το Συμβούλιο και εδώ πρέπει να πούμε ότι μάλλον βγαίνει εξασθενημένο γιατί πρέπει να συμβουδιαλέγεται με το Κοινοβούλιο και για την ε, νομοθετική διαδικασία και για τον προϋπολογισμό. Έχει έχει χάσει δηλαδή τον τελικό λόγο που είχε για τις ε, υποχρεωτικές δαπάνες. Ε, με την ε, ειδική πλειοψηφία ε, μπορούν να ληφθούν αποφάσεις πιο γρήγορα αλλά από την άλλη η δική πλειοψηφία σημαίνει επίσης ότι και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο μπορούν να προσπαθήσουν να επηρεάσουν περισσότερο τα τεκτενόμενα στο Συμβούλιο. Επομένως δεν είναι αυτό απαραίτητα ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εδώ πιστεύω ότι κερδίζει στη λήψη αποφάσεων ε, ακόμη και από την νομοθετική πλευρά, διότι με τις ρήτρε παραπομπής στα θέματα αστυνομική και δικαστικής, ε, συνεργασία, σύμφωνα με τα άρθρα της συνθήκης, προβλέπεται ε, άμεσος αντίκτυπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην νομοθετική διαδικασία. Δηλαδή, ακόμη και αν τα κράτη-μέλη ενεργοποιήσουν το μοχλό επίγουσας διαδικασίας, η νομοθετική διαδικασία κατά κάποιο τρόπο σταματά και όσο διαβουλεύεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μόνο όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαδικασία που έχει εισαχθεί, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει συνεδριάσεις επίγοντος χαρακτήρα, που σημαίνει ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μπορούν να συνεδριάσουν βάσει αυτής της διαδικασίας και να λάβουν αποφάσεις για τις τρέχουσες εξελίξεις. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε μία επιπλέον δυνατότητα για την ε, λήψη αποφάσεων που προβλέπεται για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, ε με προβλέπετε λοιπόν ε, περνάτε ήδη στην επόμενη διαφάνεια και έχουμε εδώ τις αλλαγές ισορροπίας ως προς την εφαρμογή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε αυτή την περίπτωση κάτι κερδίζει που δεν μπορεί να υποτιμηθεί τη δυνατότητα να απορρίψει τις εφαρμοστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις ε, ε, πράξεις ε, κατόπιν εξουσιοδότησης. Δηλαδή μπορεί το Κοινοβούλιο να ανασχέσει την πρόοδο κάποιων πράξεων και υπάρχει και η πλήρης συναπόφαση για τους εκτελεστικούς, τα εκτελεστικά κείμενα, τα εφαρμοστικά εκτελεστικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το ρόλο τον είχε αναγνωρίσει ατύπω το Συμβούλιο, αλλά τώρα αυτό πλέον αναγνωρίζεται και ρητά στη συνθήκη και ενισχύει το ρόλο του Κοινοβουλίου. Τώρα, η Κομισιόν έχει ενισχύσει τη θέση τη σε αυτό το σύστημα, διότι υπάρχει το σύστημα της, ε, ε, των πράξεων ε, κατόπιν εξουσιοδότησης, που περιορίζει τον έλεγχο των, της εφαρμογής από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που προβλεπόταν στις κανονιστικές και διαχειριστικές επιτροπές και κερδίζει το δικαίωμα να ξεκινήσει να ε, διαδικασίες κατά παράβαση, οπότε η Κομισιόν αποκτά μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας κατά κάποιο τρόπο και μπορεί να ξεκινήσει δυνάμει του τίτλου 6 της Συνθήκης της Λισαβόνας τις διαδικασίες κατά παράβασης, οπότε ενισχύεται κατά κάποιο τρόπο η εποπτεία της Κομισιόν. Ελπίζω ότι η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα, δεν το χρησιμοποιούσε πάντα στον τομέα των εσωτερικών ε, και ε, στον τομέα ΔΕΗ. Το Συμβούλιο είναι κάπως εξασθενημένο, διότι πρέπει να μοιραστεί τον έλεγχο που είχε πριν για τις εφαρμοστικές πράξεις της Κομισιόν. Ε, και βεβαίως ε, περιορίζεται και ο ρόλος της επιτροπολογίας με τους εμπειρογνώμονες. Οπότε το Συμβούλιο δεν έχει πλέον άμεσες εφαρμοστικές εξουσίες. Ε, που βρίσκει η θεσμική δύναμη. Το, το κοινοβούλιο ουσιαστικά δεν αλλάζει εδώ. Υπάρχουν ε, κάποιοι περιορισμοί των ε, ευρωβουλευτών, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει ουσιαστικά την ε, ισορροπία δυνάμεων. έχει αυξηθεί ο ενδοθεσμικός ρόλος της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος μπορεί να ε, υποχρεώσει κάποιους επιτρόπους να ε, ε, παραιτηθούν. Υπάρχει δηλαδή αυτή η εξουσία και σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αυξήσει τη δυνατότητα της Κομισιόν να δράσει στο εσωτερικό. Επίσης η μείωση των μελών ενισχύει κάπως τη θέση της Κομισιόν. Η βιβλιογραφία συμφωνεί ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ενίσχυση ε, στο εσωτερικό τουλάχιστον η μείωση δηλαδή των, του αριθμού των επιτρόπων. Τώρα θέτει αυτό το θέμα κατά πόσον πρέπει κάθε κράτος μέλος να εκπροσωπείται στο συλλογικό σώμα των επιτρόπων αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ανα, ε, περιορίζεται από τις παραχωρήσεις που έγιναν στην Ιρλανδία αλλά αυτό είναι εκτός ε, θέματος κατά κάποιο τρόπο, δεν, δεν το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα το Συμβούλιο ε, εξασθενεί η θέση του διότι χάνει την εκπεριτροπής προεδρία και βεβαίως υπάρχει ένα ενδεχόμενο ασυνεπιών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Ε, δηλαδή το Συμβούλιο μπορεί να χάσει στο τέλος. Υπάρχει επίσης και κίνδυνος ασυνεπιών μεταξύ του ΙΠΑ ΕΕ, του ε, προσώπου που προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών και της Προεδρίας που προεδρεύει όλων των άλλων ε, σχηματισμών. Δηλαδή έχουμε από τη μια τις εξωτερικές σχέσεις και τους άλλους, σχηματικές, ε, τους άλλους σχηματισμούς του Συμβουλίου που μπορεί να έχουν και κάποιες πτυχές που άπτονται των εξωτερικών θεμάτων και εκεί μπορεί να δημιουργήσει κάποιες ασυνέπειες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενισχύεται θεσμικά. Ήδη περιέγραψα όλες τις ε, θετικές ε, πτυχές ε, της εισαγωγής του μονίμου Προέδρου. Δεν θα μπω βέβαια σε περισσότερες λεπτομέρειες, μόνο ότι είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου το ότι μπορούν πλέον οι υπουργοί από, διάφορες ε, από τους διάφορους σχηματισμούς του Συμβουλίου να συμμετέχουν στο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αυτό ενισχύει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στους επιμέρους σχηματισμούς του Συμβουλίου. Δηλαδή μπορείς να ζητήσεις ε, σε κάποιους υπουργούς να είναι παρόντες. Θα είναι δύσκολο αυτοί οι υπουργοί στη συνέχεια να μην καταβάλουν προσπάθειες για την εφαρμογή των αποφάσεων που θα έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τέλος, η δημόσια ορατότητα. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κερδίζει θα έλεγα διότι ε, ε, η επέκταση της συναπόφασης και ε, εξουσιών ε, συγκατάθεσης ενισχύει την ορατότητα του Κοινοβουλίου. Το είδαμε και στην περίπτωση της, ε, της προσωρινής συμφωνίας SWIFT. που εμφανίζεται πλέον και στην πρώτη σελίδα των ε, εγγράφων. Ε, ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να μην χρησιμοποιεί αυτή την εξουσία αρνητικά. Αν όμως τη χρησιμοποιήσει, τελικά κερδίζει σε 42 τομείς περαιτέρω ορατότητα. Η απάντηση μπορούμε να το συζητήσουμε διμερώς αφορά ένα σχόλιο που δεν ακούστηκε από μικροφόνου. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της ενίσχυσης της ορατότητας του ε, Κοινοβουλίου η Κομισιόν κατά κάποιο τρόπο χάνει. Ε, έχουμε δύο προέδρους στην κορυφή και ήδη σε κάποια από τα ΜΜΕ μιλούν για τον κύριο Βαν Ρομπόι ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους συντομίας. Βέβαια είναι χονδροειδής απλούστευση, αλλά αυτό δείχνει την αντίληψη που υπάρχει. Και βεβαίως αυτό δεν είναι πολύ ευχάριστο για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ή, άκουσα ήδη στην ανακτήρια ομιλία του ότι θα βρει τρόπους να ε, καλύψει αυτή την πρόκληση ως προς την δημόσια εκπροσώπηση. Απλά ένα ε, σχόλιο κάνω αυτή τη στιγμή. Ε, για το Συμβούλιο Μάλλον, ε, ο ρόλος του Αντιπροέδρου και εκπροσώπου, είπα του εκπροσώπου εξωτερικών ε, θεμάτων, θα ενισχύσει το Συμβούλιο, μόνο ότι ε, η κυρία Άστον δεν αναφέρεται με το ρόλο της της αντιπροσώπου της, Ευρωπαϊκής, της αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε και εδώ βλέπουμε μία εξασθένηση του ρόλου της Κομισιόν. Η Βαρόνη Άστον αναφέρεται μόνο ως ύπατος εκπρόσωπος πολλές φορές. Οπότε ε, μάλλον το κέρδη και οι εξουσίες φαίνεται να γέρνουν προς την πλευρά του Συμβουλίου. Τώρα το Συμβούλιο ενισχύεται με το μόνιμο πρόεδρο, θα κάνει και περισσότερες άτυπες συνόδους. Ήδη ο κύριος Βαν Ρομπέι είπε ότι ζητά περισσότερες άτυπες συνόδους και ίσως το Συμβούλιο έτσι γίνει πιο ορατό. Αν τα συνδέσουμε όλα αυτά κάπως απλοϊκά, δεν έχω κάνει κάποια ποσοτική αποτίμηση. Έχω δώσει κάποια συν στους, ε, στα όργανα που κερδίζουν, μηδέν εκεί όπου δεν υπήρξε αλλαγή και μείον στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απώλεια εξουσίας και θα δείτε ότι υπάρχουν δύο νικητές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκεί έχετε την Ευρωπαϊκή, μετά έχετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο που είναι σχετική κατά κάποιο τρόπο χαμένη. Αλλά όλα είναι σχετικά. Δεν λέμε ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο τρόπο ότι έχει χάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά σε αυτό το συσχετισμό δυνάμεων είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν κερδίσει, έχουν ενισχυθεί. Ας έρθω τώρα στα συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα ε, είναι κάτι που σας παρουσίασα ήδη, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι πρωτογενής πλέον πόλη εξουσίας αυτό το ε, θεσμικό δημιούργημα, οικοδόμημα. Ε, όπως είπαμε, ε, όμως ε, εκεί βρίσκεται και η λιγότερο ορισμένη σχέση βάσει της συνθήκης. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θεσμικό κενό κατά κάποιο τρόπο. Μακροπρόθεσμα χρειάζεται να υπάρξουν στρατηγικές συμφωνίες ή συμβιβασμοί μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβίλου. Θα μπορούσε να πει κανείς ίσως και διοργανικές ρυθμίσεις ή συμφωνίας. Ο κύριος Κόρμπετ ήδη μας είπε πρόεδρος Βαν προσέφερε στο Κοινοβούλιο πιο τακτικές ενημερώσεις. Αυτό είναι ένα βήμα. Αλλά έχω τις αμφιβολίες μου κατά πόσο θα είναι αρκετό, διότι αυτοί οι δύο φορείς είναι η κύριοι πόλη του συστήματος έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα από τώρα και στο εξή. Η, η, σχετική μείωση της εξουσίας της Κομισιόν και στο νομοθετικό και στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων μπορεί να είναι ένα συμπέρασμα. Είναι σχετική αλλά αναφυσβήτητη μείωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να πιέζεται περισσότερο μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι και κύριοι ρόλοι πόλη εξουσίας και αυτό αποτελεί πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Αντιπρόεδρος Σεύκοβιτς ήδη μας είπε ότι το γνωρίζει αυτό η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι βρίσκεται σε ένα θεσμικό περιβάλλον ολοπροκλήσεις και της εύχομαι κάθε καλό αλλά είναι ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον κατά κάποιο τρόπο. Όλοι λένε ότι ο ανταγωνισμός είναι κάτι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει σας εύχομαι καλή επιτυχία. Επίσης, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως κινητήριας μηχανής ε, του συστήματος ε, αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις λόγω της ενίσχυσης του Κοινοβουλίου. Πιθανώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερο από το παρελθόν μπορεί να ε, θεωρείται ότι αυτή δεν θα είναι πλέον αυτή η οποία δίνει τις στρατηγικές απόψεις και πρωτοβουλίες διατηρεί βέβαια το ρόλο της ε, και ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει στενές συμμαχίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συμφωνία, η συμφωνία πλαίσιο ε, γιατί δημιουργεί, είναι μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει σταθερές σχέσεις με το Κοινοβούλιο ως αντίβαρο για να μπορέσει να προχωρήσει η ολοκλήρωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περιορίζει το σχετικό ρόλο του Συμβουλίου. και νιώθω τον θυμό των φίλων μου στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο είναι, μετατρέπεται σε μια σούπερ κορεπέρα, ας πούμε. Δηλαδή το Συμβούλιο προετοιμάζει τις βασικές αποφάσεις που υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το θέμα είναι τι θα γίνει, θα έχουμε ένα senior και ένα junior κορεπέρ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά λέω να η τάση είναι να περιοριστεί σχετικά η θέση του Συμβουλίου. Η νέα θέση του είπα του εκπροσώπου αντιπροέδρου είναι ένα περίεργο δημιούργημα, ίσως ε, τα μοναδικά περίεργα ε, δημιουργήματα. Ε, υπάρχουν βέβαια νομικές, πολιτικές, έτσι περίεργες οντότητες, αλλά οι διαπραγματευτές δημιούργησαν κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ αλλά ε, δεν έχει ακόμα επαρκή δημοκρατική κατά κάποιο τρόπο νομιμοποίηση μέσα σε αυτό το τρίγωνο. Και είναι δύσκολη η θέση και η δουλειά θα έλεγα. Ίσως η πιο δύσκολη θα έλεγα εγώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είμαι 100% αισιόδοξο ε, για την μακροβιότητα και μακροπρόθεσμη σταθερότητα της επισφαλούς αυτής θέσης. Άρα πρέπει να την παρακολουθήσουμε. Η επιπλέον πολυπλοκότητα τώρα και οι αλλαγές στην ισορροπία σχέσεων ε, κάνουν τις ε, οργανικές διαρρυθμίσεις ε, πιο απαραίτητες από ποτέ. Το σύστημα δεν θα προχωρήσει εάν δεν επιτυγχάνει συμβιβασμούς για να υπάρχει ροή πληροφοριών και σχέσεις εμπιστοσύνης. Δηλαδή μέσα από συνθήκες, συμφωνίες, συνεδριάσεις Χρειάζεται περισσότερο από ποτέ διοργανική συνεργασία. Το σύστημα πιθανώς να μην λειτουργήσει εάν δεν το διαχειριστούμε σωστά. Και εδώ κύριε Αντιπρόεδρε έχετε βαριά ευθύνη. Τέλος, τελική διαφάνεια στην ε, πολιτική πράξη ή στον ακαδημαϊκό χώρο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ε, ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει αλλά πρέπει να θυμίσουμε το βιβλίο του, της βίβλου Δανίλη 527 που ε, λέει ότι ζυγίζεστε στη ζυγαριά και βρίσκεστε να υπολείπεστε. Η βίβλος λέει πολλές φορές πολύ ε, φρικτά πράγματα για την πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μονάρ. Η κυρία Λουτσία Σερένα Ρώση. Ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου που είμαι ανάμεσά σας. Έχω και εγώ παρουσίαση PowerPoint, αλλά μόνο ελάχιστες διαφάνειες θα δείξω, γιατί έχουν ήδη ε, με έχουν ήδη καλύψει προλαλήσαντε. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον καθηγητή Μόναρ και τη δική του ανάλυση των πραγμάτων. Εγώ εξετάζω θέματα παγκόσμιων ισορροπιών. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάλλον πιο υπερεθνική ή πιο διακυβερνητική μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό εξετάζω. Ποια είναι η κατεύθυνση προς την οποία οδεύει το όλο σύστημα, ποιες ε, εξελίξεις αναμένονται βλέπετε εδώ πέρα παρήθμιση θεσμικών οργάνων. Δεν λέω ότι το, η υπερεθνική διάσταση ε, αντίκειται στη διακυβερνητική. Να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Η Κομισιόν ήταν στο επίκεντρο της κοινοτικής μεθόδου, ήταν ο, ο θεματοφύλακας της, ε, του υπερεθνικού χαρακτήρα του συστήματος, ενώ το Συμβούλιο πίεζε προς μία πιο διακυβερνητική εξέλιξη. Τώρα φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ενισχυθεί καθοδόν και αποτελεί πλέον ένα παράγοντα της υπερεθνικής ε, κατεύθυνσης. Και υπάρχει βεβαίως και το ΔΕΚ που καταρχήν θα πρέπει να είναι αμερόληπτο βεβαίως και να κρίνει αλλά το δικαστήριο, πώς να το κάνουμε, έχει το δικό του όραμα περί Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμφισβήτητα και πρόκειται για υπερεθνικό όραμα. Οπότε έχω βάλει στην, ε, στα αριστερά, στην υπερεθνική στήλη, Κομισιόν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ΔΕΚ. Και στην άλλη στήλη, διακυβερνητική κατεύθυνση, έβαλα το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρθρο 10 τη συνθήκη έχει προβλέψει την κυβερνητική διάσταση με αυτή την ε, διτή δομή. Ας ε, πάρουμε ξεχωριστά το κάθε θεσμικό όργανο. Πράγματι το Συμβούλιο σαφώς και έχει ενισχυθεί. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σαφώς και έχει ενισχυθεί από τη συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αυτός που πραγματικά χαράσει η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δίνει τη γενική πολιτική κατεύθυνση, ε, χαράσει τις προτεραιότητες, ε, τους στόχους ακόμα της εξωτερικής δράσης και το καθεξής. Μετά έχουμε τη θεσμική έκπληξη που είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γιατί αποτελεί έκπληξη αυτός ο άνθρωπος Διαβάζοντα τη συνταγματική συνθήκη, μετά και προ και μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα, θα μπορούσε κανεί να φανταστεί ότι ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ήταν απλά ένα υπερεθνικό γραμματέα. Ε, ενώ σε σχέση με τη δομή αυτή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. Αλλά στην πράξη μας κατέπληξε ο κύριος Βαρόμπόη, διότι αναλαμβάνει ενεργό ρόλο με ετήσιες σχεδόν ε, συνόδους, ε, με πολλές ε, συνόδους, με πολλές επαφές διεθνείς του κυρίου Βανοπόη και μπορεί να αναμένεται ακόμα μεγαλύτερος ρόλος κατά την, με την επερχόμενη προεδρία τη Βελγική. Ο κύριος Βαρομπόη θα ακόμα πιο ελεύθερα θα παίξει ενισχυμένο ρόλο με την επερχόμενη Βελική Προεδρία. Να δούμε το Συμβούλιο. Αποδυναμώνεται, εξασθενεί ο ρόλος του. Λόγω του ενισχυμένου ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα απλά εκτελεί πλέον τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις προτεραιότητές του είναι αναγκασμένο να μοιράζει τις νομοθετικές του εξουσίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλο και περισσότερο. Τώρα, οι νέοι κανόνες ε, περί εξουσιοδότησης και εκτέλεσης, ενδεχομένως κατάργηση επιτροπολογίας, Αποδυναμώνεται λοιπόν το Συμβούλιο και πλέον δουλεύει επίσης όρες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, οι σχηματισμοί του Συμβουλίου έχουν αλλάξει τα πράγματα εκεί πέρα ως προς την ε, Προεδρία τους. Υπάρχει ίσως κάποιο πρόβλημα ορατότητας ε, του Συμβουλίου ως ε, θεσμικό όργανο πάντα. Και κάτι ακόμα. Ο ρόλος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων φαίνεται πολύ αβέβαιος. Δεν είναι σαφές ποιος εποπτεύει την εγκάρσια συνοχή των επιμέρους σχηματισμών του Συμβουλίου. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Συμβούλιο Γενικών ε, Υποθέσεων, ε, τη συνοχή στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων την διασφαλίζει η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων. Άρα και ο ρόλος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων έχει εξασθενήσει μετά, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον έχει ενισχυμένε εξουσίε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περισσότερε νομοθετικέ εξουσίε, δουλεύει πλέον επίση όροι σε θέματα εξουσιοδότηση με το Συμβούλιο, μεγαλύτερε δημοσιονομικέ εξουσίε, μεγαλύτερη υποπτία των άλλων θεσμικών οργάνων και αυξανόμενη πολιτική επιρροή. Στα γρήγορα μπορούμε να δούμε τι επόμενε διαφάνειες, γιατί όλα αυτά έχουν ήδη υποθεί, περισσότερες νομοθετικέ εξουσίες, αλίμονο και όχι μόνο στην απόφαση που έχει αυξηθεί και καλύπτει ως και το 90% του νομοθετικού έργου έχει και το δικαίωμα πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναθεώρηση της συνθήκης. αλλά έχει κάθε δυνατότητα να στραφεί στην Κομισιόν και να, να απαιτήσει την κατάθεση από πλευρά Κομισιόν ε, προτάσεων. Την εξουσιοδότηση την ανέφερα. Μετά, επέκταση και τη συγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διαγράφεται μια ενδιαφέρουσα τάση κατά τη γνώμη μου. Προηγουμένω τη συγκατάσταση την αποκαλούσαμε συνένεση. Και ήταν ένα είδο εκ των ελέγχου. Ήταν σαν, σαν ένα πυρηνικό όπλο, α πούμε, ε, που θα ήταν υπερβολικές οι ζημίες του για να χρησιμοποιηθεί. Ας πούμε, σε θέματα ένταξης νέων κρατών μελών δεν ε, το αξιοποιούσαμε γιατί, θεωρούνταν, ε, γιατί θεωρούσαμε υπερβολικέ τι συνέπειε. Όμω στην πράξη τι έχουμε δει, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιοποιεί και αυτή την εξουσία και αυτή τη δυνατότητα τη συγκατάθεση που σαφώ και έχει επεκταθεί σε κάποιους νέου τομεί με τη Λισαβόνα με τρόπο προληπτικό, εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων πλέον. Διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να επηρεάσει ε, πράγματα και καταστάσεις. Και γι' αυτό δεν παρέχει τη συγκατάθεσή του σε κάποιες περιπτώσεις. Και με αυτόν τον τρόπο ασκεί επιρροή το Κοινοβούλιο σε σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα. Ε, ασκεί αυτή την εξουσία με τρόπο προληπτικό. Περνάμε στις δημοσιονομικές εξουσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυξημένες, ενισχυμένες δημοσιονομικές ε, εξουσίες στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΕΠΑ και σε πλαίσιο εξωτερικών σχέσεων, δείτε ας πούμε την όλη συζήτηση για την ε, Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Υπηρεσία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιοποιήσει αυτές τις δημοσιονομικές του εξουσίες ε, για να επηρεάσει, για να ασκήσει επιρροή σε θέματα εξωτερικής διάστασης, σε θέματα ΚΕΠΑ, όπου ο συνομοθέτης δεν διαθέτει αρμοδιότητες πάμε στις εποπτικές εξουσίες, εξουσίες ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάλι ενισχύθηκαν. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε οι εξελίξεις στι σχέσεις μεταξύ Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μαθητής της Κομισιόν. Υπό την αιγίδα της Κομισιόν. Θυμάστε την ε, περίφημη υπόθεση ε, όταν και στράφηκε το Ευρωκοινοβούλιο ενώπιον του ΔΕΚ με τη βοήθεια της Κομισιόν σε θέματα που αφορούσαν νομικέ βάσει. Αλλά μετά από κάποια χρόνια αντιστράφησαν ε, οι ρόλοι. Το είδαμε σαφώς και με την πρώτη και με τη δεύτερη κομισιόν. Το βλέπουμε σαφώς και με την πρώτη και με τη δεύτερη κομισιόν Παρόσο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι που έχει λόγο σε σχέση με τη σύνθεση της Κομισιόν. PNR, SWIFT, ACTA, είχαμε όλα αυτά τα παραδείγματα ε, σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες και την παραχάραξη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έπαιξε ενεργό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η ειδική σύμπραξη, η ειδική εταιρική σχέση. Χάρη στη νέα συμφωνία πλαίσιο που διαπραγματεύτηκε ο κ. Σκόρμπετ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η νέα διοργανική συμφωνία, πράγματι. διότι μιλάμε πλέον για νέες σχέσεις με την Κομισιόν που οφείλει να ενημερώνει, να προσκαλεί στις εργασίες της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί το Κοινοβούλιο να εξαργάσει την Κομισιόν σε επιμέρους απολύσεις και η διοργανωτική συμφωνία προβλέπει μεγάλο συντονισμό, συνεχή ενημέρωση και νέες ισορροπίες στις σχέσεις Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμα και σε θέματα διαπραγμάτευσης διεθνών συμφωνιών. Εξαστε... Αποδυναμωμένη Κομισιόν πιθανότατα ναι. Έχουμε αποδυναμωμένη πράγματι Κομισιόν με την... υπό την παραδοσιακή έννοια του όρου αλλά η Κομισιόν αλλάζει πάντως ρόλο. Και εδώ πέρα δεν είναι θέμα στάθμισης επιμέρους εξωσιών. Αλλάζει ρόλο η Κομισιόν. Τώρα η Κομισιόν ευθύνει πιο διακυβερνητική προσέγγιση. Λόγω και της σύνθεσης της Κομισιόν. Διότι με 27 επιτρόπους μόνο αυτό είναι εφικτό. Καμιά φορά οι επίτροποι, πώς θα το κάνουμε, εκπροσωπούν εθνικά συμφέροντα. Θα πρέπει να περιοριστεί η σύνθεση της Κομισιόν, αλλά υπάρχουν ε, μεγάλες ε, αντιρρήσεις από το 2014 και μετά. Υπάρχει πολιτική συμφωνία να μην περιοριστεί η σύνθεση της Κομισιόν. Μόνο με ομοφωνία μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Περιορίζονται πάντω οι προτάσει από πλευρά Κομισιόν. Παρουσιάζει όλο και λιγότερο λιγότερες προτάσεις Κομισιόν σε θέματα ιδίως ε, ΔΕΗ. Οι προτάσεις θα πρέπει να προέρχονται από ένα τέταρτο των κρατών μελών σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά βεβαίω τα κράτη-μέλη δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να παρουσιάσουν προτάσεις. Περιορίζονται στον αριθμό οι προτάσεις λοιπόν της Κομισιόν. Και το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι χάνει πολιτική όθηση η Κομισιόν, διότι το ρόλο αυτό τώρα τον αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο νέο σύστημα. Οπότε, αν συγκρίνουμε τούτη εδώ την Κομισιόν με την προηγούμενη, με με την Κομισιόν Τελόρ, τι βλέπουμε, ότι τη στιγμή του Τελόρ την πολιτική όθηση σαφώς και την έδωνε η Κομισιόν. Με τις προτάσεις της. Προτάσει τη που ήταν στρατηγικέ προτάσει ενώ τώρα τη στρατηγική τη χαράσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που επηρεάζεται όλο και περισσότερο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν ε, είναι που εφαρμόζει στην πράξη τη στρατηγική που χαράσεται σε άλλο επίπεδο. Δεν ξέρω κατά πόσον έχει αποδυναμωθεί η Κομισιόν, πάντως η Κομισιόν αλλάζει. Αλλάζει ρόλο. μπορεί να θεωρηθεί και φυσικό βεβαίως. Είναι η φυσική εξέλιξη ας πούμε του συστήματος. Βεβαίω θα πρέπει να πετύχουμε σωστέ ισορροπίε για να μην χαθεί η κοινοτική υπερεθνική μέθοδο. Όλα αυτά θα τα αναφέρω στο τέλο τη παρουσίασή μου. Τώρα θα πάμε ακόμα πιο γρήγορα. Περνάμε στον ύπατο εκπρόσωπο σε θέματα ΚΕΠΑ. Ιδού άλλη μία αποστολή της ΥΠΑ του εκπροσώπου. Είναι σκληρή δουλειά. Το θέμα είναι ποιος μιλάει με τη μία φωνή της ε, Ένωσης. Δείτε τι γίνεται σε επίπεδο ΟΙΕ. Δεν είναι καθόλου εύκολο να υπάρχει ορατότητα και κοινή εκπροσώπηση της Κομισιόν. Ορθά και δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μου η Κομισιόν ε, δεν δέχεται αυτά που λέει το Συμβούλιο προκειμένου. Τώρα τι διακυβεύεται στην περίπτωση Mercury. Είναι ισορροπίες μεταξύ Κομισιόν και Συμβουλίου στην περίπτωση μεικτών συμφωνιών. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Άλλο σύμπτωμα τώρα του νέου αποδυναμωμένου διαφορετικού τέλο πάντων ρόλου της Κομισιόν είναι το λεγόμενο gentrification. Παχάρου από 40 είναι κοινοτικοί οργανισμοί αυτή τη στιγμή. Παίζουν ρόλο που παλιά τον έπαιζε η Κομισιόν. Είναι μεγάλος ο έλεγχος βεβαίως σε αυτούς τους κοινοτικούς οργανισμούς ε, εκ των υστέρων βεβαίως κυρίως από το δικαστήριο, από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ας πούμε σε σχέση με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι το ψήφισμα περί συμφωνιών πλαίσιο ζητάει και κοινοβουλευτικό έλεγχο για τους εκτελεστικούς διευθυντές σε αυτούς τους οργανισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι μεν αυτόνομοι, αλλά όχι και υπερβολικά αυτόνομοι. Τώρα, να δούμε το ΔΕΚ. Αλλή μόνο. Οπωσδήποτε θα πρέπει να το καλύψουμε και το ΔΕΚ. Επίσης έχει ενισχυμένες εξουσίες. Γιατί πλέον έχει δικαιοδοσία σε πράξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όταν ψηφίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, στους οργανισμούς της Ένωσης σε σχέση με την ε, αναθεώρηση νομιμότητας και για τα προδικαστικά ερωτήματα, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους κοινωτικούς οργανισμούς. Διότι οι κοινοτικοί οργανισμοί έχουν επαφές με τους πολίτες. Άρα τα προδικαστικά ερωτήματα είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πολύ χρήσιμη αποστολή του ΔΕΚ. Παίζει συνταγματικό ρόλο το ΔΕΚ και αυτό είναι αποτελεί απόρρια της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το ΔΕΚ χρειάστηκε να υπεραμεινθεί των θέσεών του και εν ώψη της ε, συνέλευσης, Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το ΔΕΚ ε, όλο και περισσότερο βασίζεται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το δικαστήριο τελικά είναι ο τελευταίος διαμεσολαβητής σε αυτό το σύστημα. Δεν νομίζω να, αλλάξει, να αλλάξουν κατεύθυνση. Τώρα, ποιε είναι οι νέε ισορροπίε που έχουν διαμορφωθεί. Είναι πιο υπερεθνική ή πιο διακυβερνητική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν απλά δούμε τις επιμέρους εξουσίες του κάθε θεσμικού οργάνου μπορούμε να πούμε ότι στην υπεραθνική διάσταση αυτά που έχασε η Κομισιόν τα κέρδισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις απώλειες του Συμβουλίου τις αντισταθμίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα είναι μηδενικό το αποτέλεσμα μεταξύ ε, υπερεθνικής και διακυβερνητικής ε, διάστασης. Παραμένουν ε, οι ίδιες ισορροπίες. Αλλά στην πράξη αυτό δεν αληθεύει και τόσο. Διότι ε, το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι δυνατό να δώσει την πρωτοκαθεδρία στη διακυβερνητική πλευρά. Λόγω του ισχυρότατου ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ελοχεύουν κίνδυνοι. Διότι σε πλαίσιο διακυβερνητικό οι συμβιβασμοί βεβαίως και είναι απαραίτητοι, ενώ τώρα θα πρέπει να νοιαστούμε για το γενικό συμφέρον παραπόλα. Επόμενη διαφάνεια. Αλλάζει ο ρόλος της Κομισιόν. Πολύ προκλητικά αυτά που λέω στη διαφάνεια μου βεβαίως. Υπέργραμματεία του Συμβουλίου, η τμήμα μελετών ελοχεύουν ε, αυτοί οι κίνδυνοι εάν ε, η Κομισιόν δεν προχωρήσει σε σύμπραξη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε συμμαχία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυκλοφορούν κάποιες ιδέες ε, με τις οποίες δεν συμφωνώ απαραίτητο, ας πούμε συγχώνευση μεταξύ των Προέδρων της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν συμφωνώ, αλλά κάποια think tanks προωθούν τέτοιες ιδέες άμεση εκλογή του Προέδρου της Κομισιόν. Από το BVG στην Λισαβόνα, εκεί πέρα κυκλοφορούν αυτές οι ιδέες. Δεν είναι κακή ιδέα. Αλλά στην πράξη δεν το βλέπω και τόσο εφικτό παρότι θα ενίσχυε τη δημοκρατική νομιμότητα της ε, Κομισιόν. Θα χρειαζόταν τροποποίηση και πάλι της συνθήκης. Κατά την επόμενη εκλογή του Πρόεδρου της Κομισιόν θα ήταν χρήσιμο τουλάχιστον κάθε πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρουσιάσει έστω το δικό της υποψήφιο. Αυτό θα σήμαινε ενισχυμένο έλεγχο της Κομισιόν και ενισχυμένη ορατότητα για τον πρόεδρο της Κομισιόν. Άρα, πώ πετυχαίνουμε τις λεπτές ισορροπίες σε αυτό το σύστημα. Το πρώτο Κοινοβούλιο έχει να παίξει ρόλο στο η μελλοντική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τώρα, ένα διαφορετικό σενάριο ποιο θα ήταν. Όχι ακριβώς συντονισμός, που ήδη ακούστηκε μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά τουλάχιστον ε, συνεχής διάλογος ε, μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με ισχυρό πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μοιράζεται μόνο το νομοθετικό ρόλο με το Συμβούλιο, αλλά και την πολιτική όθηση και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εδώ και χρόνια γίνεται λόγος για δημοκρατικό έλλειμμα. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος του προβλήματος, διότι η συναπόφαση πλέον έχει επεκταθεί και φτάνει και το 90% ε, της νομοθετικής διαδικασίας. Το θέμα είναι το πολιτικό έλλειμμα. Γιατί δεν έχουμε ακριβώς υπερεθνικά κόμματα. Άρα αυτό είναι ο μελλοντικό στόχος. Να καλύψουμε αυτό το χάσμα, αυτό το πολιτικό έλλειμμα. Αυτό θα πρέπει να είναι η μελλοντική στόχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν χρειάζεται περισσότερε εξουσίε. Νέο όραμα τη Ευρώπη χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπου θα πρωτοπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ ονόματο ε, των Ευρωπαίων πολιτών, ένα κοινοβούλιο που θα βασίζεται στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στα ένδικα μέσα, στην πολιτική επιρροή και μάλιστα με τρόπο ιδιαίτερα ενεργό. Πράγματι το κοινοβούλιο είναι μαχητικό. Ε, το έχουμε δει πρόσφατα στο μέτωπο των διεθνών συμφωνιών. Θα πρέπει πλέον να μιλάμε για υπερεθνικά κόμματα, υπερεθνικές εκστρατείες, υπερεθνικές αξίες. Μόνο έτσι πετυχαίνουμε τις σωστές ισορροπίες ε, και πετυχαίνουμε την μετάβαση στην διακυβερνητική μέθοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρώση. Νομίζω ότι η πανεπιστημιακή διάσταση διεύρυνε την αμυγός πολιτική διάσταση στη συνεδρία αυτή. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως τη συζήτηση. Δεν ξέρω πόσο... Πέντε λεπτά να αφήσω για τη συζήτηση. Ξέχασα, συγγνώμη, ξέχασα, συγγνώμη, συγγνώμη σας, ξέχασα. Χίλια συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Μ' ακούτε? Θα μιλήσω γαλλικά. Όπως ξέρετε, γιατί αν δεν το ξέρετε θα σας το εξηγήσω, είμαι δημοσιογράφος εγώ δεν έχω τίποτα το επίσημο, μιλώ εξ ονόματός μου προσωπικά και η οπτική μου είναι εντελώς διαφορετική από αυτή των ομιλητών που μίλησαν υπό την έννοια δηλαδή ότι εγώ είμαι χρήστης των θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Οπότε θα σας πω πώς λειτουργούν από την πλευρά όπως τις βλέπουν δηλαδή οι χρήστες. Πρώτα πρώτα θα έλεγα ότι το σπουδαίο με τις ε, καινοτομίε που ήδη άρχισαν εν μέρη να ισχύουν, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποιες αβεβαιότητες, κάποιες ασάφειες και το βλέπω στην καθημερινή μας δουλειά των ε, δημοσιογράφων ε, του πρακτορείου Agence Europe και το ζούμε καθημερινά. Οι δύο σημαντικές, οι δύο βασικές πτυχές είναι πλέον ξεκάθαρες για μας και για τη δουλειά μας. Η πρώτη πτυχή αφορά τη νέα εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συν νομοθέτη που εμπλέκεται άμεσα σε τομείς από τους οποίους ήταν, ε, αποκλειόταν στο, στο, στο παρελθόν ε, παρά μόνο όταν επρόκειτο να μιλήσει όχι στη, δεν συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων όπως ήταν η εμπορική πολιτική και η γεωργία. Βλέπουμε λοιπόν πως η νέα εξουσία του Κοινοβουλίου ε, τροποποιεί τη λειτουργία της Ευρώπης. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, θα μπορέσουμε να επανέλθουμε αν τεθούν συγκεκριμένα ερωτήματα. Η δεύτερη πτυχή μετά από αυτή του Κοινοβουλίου, ε, που είναι σαφής για τη λειτουργία της πλέον, είναι η τροποποίηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον ε, μόνιμο Πρόεδρο κλπ. Κατά τη γνώμη μου, όλα τα οποία συνέβησαν σε αυτή τη μεταρρύθμιση είναι γενικώ θετικά μολονότι θα μπορούσε να κάνει κανείς κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις. Στον τύπο ε, επικρίθηκε η επιλογή του μονίμου Προέδρου, διότι κατά ορισμένους ε, δημοσιογράφους δεν ήταν τόσο γνωστός στην κοινή γνώμη, ε, στον κόσμο ή στην Ευρώπη. Υπήρξαν δημοσιεύματα που τον ανέφεραν ως Mr. Nobody, ο κύριος κανείς για να τον κατονομάσουν. Κατά τη γνώμη μου είναι σφάλμα αυτό. Ε, ένας γνωστός, μια γνωστή προσωπικότητα θα είχε ε, έρθει με τις πεπιθήσεις του, με το παρελθόν του και θα είχε ουσιαστικά πολύ περισσότερες δυσκολίες. Ο κύριος Βανορομπέη δεν το προφέρω σωστά, αλλά καταλαβαίνετε τώρα για ποιον μιλώ ξεκίνησε ε, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του και έκανε μία δήλωση πολύ μετριοπαθή αλλά μάλλον έτσι ευστοχή και έξυπνη και σημαντική. Ε, είπε οι προσωπικές μου ε, απόψεις δεν έχουν καμία σημασία. Δεν θα τις εκφράσω ποτέ. Οι θέσεις που θα υποστηρίξω ενώπιον της κοινή γνώμης του τύπου κλπ θα είναι οι θέσεις του ε, τη Συνόδου Κορυφής συνολικά. Εκ πρώτης όψεως αυτή η δήλωση ε, εξέφραζε με τριοπάθεια. Στην πραγματικότητα όμως σήμαινε τι δίνω ε, σπουδαιότητα σε αυτά τα οποία λέω. Δηλαδή οποιαδήποτε λήψη από ε, θέσεις από πλευράς του κυρίου Βαν Ρομπέη είναι οι θέσεις του Συμβουλίου. Οπότε καταλαβαίνετε το βάρος που έχει η κάθε διακήρυξη. Οπότε βεβαίως καταλαβαίνετε με πόση προσοχή τον παρακολουθούμε εμείς. Το γεγονός ότι δεν ήταν γνωστό στο παρελθόν δεν έχει πια καμία σημασία και είχε τη δυνατότητα να κάνει και κάποιες σημαντικές δηλώσεις, θα έλεγα σχεδόν επαναστατικές, όταν είπε ότι η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης, η οικονομική κυβέρνηση της Ευρώπης υπάρχει και είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και προσέθεσε και δύο προτάσεις για να εξηγήσει γιατί. Είναι πολύ προσεκτικός στους όρους που χρησιμοποιεί και δεν θέλει να μπει στη διαμάχη ευρωπαϊκή κυβέρνηση, ευρωπαϊκή διακυβέρνηση που αλλάζει ανάλογα με τη γλώσσα. Το σημαντικό για μάλλον για αυτόν είναι και τα δύο. Είτε το πούμε διακυβέρνηση είτε το πούμε κυβέρνηση είναι κάτι που υπάρχει. Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε κάτι καινούργιο και είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εξάλλου ε, η λέξη κυβερνητικός προκύπτει από το γεγονός ότι στην πράξη ο κύριος Βανρομπέ συγκαλεί τη συνοδοκορυφή σχεδόν κάθε μήνα. Ε, κάνει μια συνεδρίαση, εξηγεί για ποιο λόγο, με ποιο θέμα, ε, σε τι θα εστιάσει την προσοχή της. Και το ίδιο ισχύει και για την προετοιμασία. Αλλά στην ουσία όταν έρχονται οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μιλούν για όλα τα θέματα της επικαιρότητα και ε, συζητούν για τα πάντα. Η τρίτη επανάσταση, θα λέγα η επανάσταση η οποία προκύπτει από αυτή τη συνεχή σύγκληση, σημαίνει συμμετοχή, άμεση συμμετοχή, μόνιμη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ίσως ακούγεται κοινότυπο, θα μου πείτε είναι φυσιολογικό να ασχολούνται οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων με την Ευρώπη, αλλά αυτό δεν ίσχυε πριν. Υπήρχαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που είχαν κάποια αόριστη γνώση, κάπως έτσι αφηρημένα και επιφανειακά γνώριζαν τα ευρωπαϊκά πράγματα. Για ορισμένους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το ουσιαστικό στοιχείο του εξαμήνου της Προεδρίας τους ήταν να συναντούν τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε. Κατηδίαν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μου είπε ότι συχνά η, η, βοηθή του προέδρου της, ε, των Ήπα πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, ρωτούσαν «Μα ποιος είναι τούτος εδώ, δεν ξέραν από πού προερχόταν καν». Ε, πήγαινε για μερικές μέρες και μετά, ξέρω εγώ, ένα μήνα μετά, δύο μήνες μετά δεν ήταν πλέον πρόεδρος και ε, βρισκόμασταν σε μία κατάσταση όπου η υπερευαισθησία ορισμένων, η ευθυξία ορισμένων ε, μπορούσε να υποστεί πλήγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι γενικώ είναι καλό για την Ευρώπη το ότι έχουμε μόνιμο πρόεδρο. Μετά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάποιο παρατήρησε ότι κανένα δεν είχε μιλήσει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τύπο τόσο όσο αυτή τη στιγμή. Οι δημοσιογράφοι βεβαίως κατάλαβαν τι είναι το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο ε, αποφασίζει, συναπόφαση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η θεσμική λοιπόν μετατροπή της, της Ευρώπης είναι κάτι ζωντανό. Για κάποιες άλλες πτυχές δεν έχω ακόμα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, θα πρέπει να δούμε στην πορεία, στην πράξη. Ε, ε, αυτό ισχύει κυρίως ε, για τους υπευθύνους της διπλωματικής υπηρεσίας που είναι ύπατος εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη, ομολογώ ότι για μας τους δημοσιογράφους δεν είναι και ξεκάθαρο απόλυτα. Νομίζω ότι το βασικό, η βασική αμφισημία κατά κάποιο τρόπο στον τύπο και έχει άδικο ο τύπος είναι να παρουσιάζει την ε, κυρία που εκπροσωπεί αυτή τη θέση ως Ευρωπαίο Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό είναι ε, λάθος ονομασία η οποία ε, ουσιαστικά παραπλανεί τη γνώμη. Δεν υπάρχει ακόμα ευρωπαϊκή πολιτική εξωτερικών. Εξάλλου και ο πρόεδρος είχε κάνει μια πρόταση, μια δήλωση για αυτό το θέμα. Για την ώρα το καθήκον της θέσης αυτής, της υπηρεσίας αυτής και του ατόμου που βρίσκεται επικεφαλής είναι να συμβάλλει στη δημιουργία μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής εξωτερικών που θα έρθει κάποια στιγμή, τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε, αρχίζουμε να συζητάμε μαζί για τα προβλήματα. Αλλά είναι σφάλμα αυτή τη στιγμή να μιλούμε για υπουργό εξωτερικών και για πλειοψηφική ψήφο για να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο θέμα της πλειοψηφίας. Θα ήθελα να σας δώσω δύο παραδείγματα για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Ένα παλιό παράδειγμα και ένα σύγχρονο. Από τις αναμνήσεις μου ανασύρω ένα παράδειγμα την εποχή που ξέσπασε ο πόλεμος του Ιράκ. Τότε είχε συνεδριάσει η ε, ε, Σύνοδος για να συζητήσει την κοινή πολιτική ασφάλειας και εξωτερική πολιτική. Οπότε τότε υπήρξε η ρήξη μεταξύ των κρατών μελών που συμμετούχαν στον πόλεμο και των κρατών που δεν ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτό τον πόλεμο. Υπήρξαν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι είπαν «Μα τι κάνουμε» δεν έχουμε ακόμα κανόνες ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας και τα σπάσαμε όλα. Ε, μεγάλη ζημιά πραγματική και τότε δύο προσωπικότητες τις οποίες θα κατονομάσω, ένας ήταν ο Ζακ Ντολόρ και ο άλλος ήταν ο Ζης Καρδεστά που ήταν ε, πρόεδροι της συνόδου αυτής, μου είπαν ξεχωριστά ο καθένας, αλλά κατ' ουσίαν το ίδιο. Αν είχαμε τότε, τότε την ε, ΚΕΠΑ με πλειοψηφική ψήφο θα είχαμε σπάσει την Ευρώπη στα δύο. Διότι ποτέ τότε το Ηνωμένο Βασίλειο και κάποια άλλα κράτη-μέλη της Αναταλικής Ευρώπης δεν θα είχαν δεχτεί να παρετηθούν από τη συμμετοχή τους από τον πόλεμο αυτό και το άλλο μέρος της Ευρώπης με επικεφαλής Γερμανία και Γαλλία θα είχαν δεχτεί να ε, συμμετα... δεν θα είχαν δεχτεί να συμμετάσχουν. Το αποτέλεσμα της ψήφου δεν θα ήταν τόσο σημαντικό. Αν είχαμε ε, μπορέσει να ψηφίσουμε και να πούμε έχουμε κοινή πολιτική και ψηφίζουμε τώρα, θα είχαμε σπάσει την κοινή πολιτική, την κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρώπης στα δύο. Σας είπα λοιπόν ότι θα σας έδινε δύο παραδείγματα. Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο είναι ένα επίκαιρο με θέμα το Κόσοβο. Ίσως ξέρετε ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνώρισε το κοσυφοπαίδιο. Υπάρχουν κράτη-μέλη που το αναγνώρισαν και κάποια κράτη-μέλη που δεν το αναγνώρισαν. Και πάλι, αν έπρεπε να πούμε υπάρχει εξωτερική πολιτική, άρα ψηφίζουμε, και πάλι θα είχαμε προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες στην Ευρώπη, γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι λόγοι για τους οποίους κυρίως η Ισπανία δεν αναγνώρισε το κοσυφοπέριο έχουν κάποια σημασία. έχουν σημασία όχι για το κοσυφοπέδιο ε, αυτό καθ' αυτό είναι ένα πρόβλημα μπορεί να επιληθεί αλλά διότι θα σήμαινε από νομική απόψεως ότι δεχόμαστε την αρχή ότι μια χώρα του ΟΗΕ η μέρος αυτής της χώρας μπορεί να αποσχιστεί και να κηρύξει την ανεξαρτησία του ε, χωρίς να υπάρχει συνένεση συνολικά της χώρας. Ε, και μια χώρα όπως η Ισπανία που έχει το πρόβλημα της χώρας των Βάσκων και κάποιες αποσχιστικές τάσεις της Καταλωνίας όπως ισχυρίζονται ορισμένοι δεν θα μπορούσε να δεχτεί να, να, να γίνει δυνατόν και να σας πω για ποιο λόγο. Γι' αυτό το λόγο είπε όχι. Η ευρωπαϊκή πολιτική, κοινή πολιτική δεν υπάρχει, δεν υπάρχει Ευρωπαίος Υπουργός Εξωτερικών έτσι πρέπει να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Και έτσι θα το κάνουμε και στα πλαίσια της δουλειάς μου. Τελείωσα κύριε Πρόεδρε. Το τελευταίο που θέλω να πω αφορά τις ενισχυμένες συνεργασίες. Υπάρχουν πολλοί που δεν πιστεύουν ότι η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει με 27 κράτη-μέλη. Μπορεί ναι, να προχωρήσει συνολικά, αλλά δεν μπορεί να υλοποιήσει ορισμένα πράγματα ε, με 27 μέλη. Και το μέσο της ενισχυμένης συνεργασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Και δεν μιλώ θεωρητικά, διότι δεν είναι ο ρόλος μου, δεν είμαι καθηγητής πανεπιστημίου. Εγώ το λέω πώς λειτουργεί στην πράξη. Η πρόταση του Ζακ Ντολόρ, όχι μόνο του δηλαδή, αλλά ήταν επικεφαλής μιας ομάδας να δημιουργηθεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και είχε πει δεν είναι δυνατόν, υπάρχουν χώρε που δεν συμφωνούν, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την οδό της ενισχυμένης συνεργασίας. Δηλαδή τα κράτη που θέλουν να συμμετάσχουν συμμετέχουν και όσοι δεν θέλουν μπορούν να συμμετάσχουν αργότερα. Βέβαια το θέμα είναι πολύ λεπτό, το ξέρουμε αυτό. Οι χώρες που είναι στο περιθώριο φοβούνται μήπως η Ευρώπη χωριστεί στα δύο, σε δύο σειρέ πρώτης κατηγορίας και δεύτερη κατηγορία. Ο Ζακ Ντολόρ λοιπόν εφήβρε μια λέξη που όπως είπε ο ίδιο δεν του πολύ αρέσει, αλλά μίλησε για τη διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση, που είναι εύσχημος τρόπος για να μην ε, ε, θίξει τις ευαισθησίες των χωρών εκείνων που για την ώρα δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε νέα πρωτοβουλία, αλλά παρά όλα αυτά χρειάζονται κάποιες νέες πρωτοβουλίες και δεν χρειάζεται, δεν μπορούμε να τα σταματάμε όλα. Ο Ντελόρ υποστηρίζει με διαφορετικό ίσως τρόπο όχι αυτό τον που έχουν οι ενισχυμένες συνεργασίες, αλλά με διαφορετικές μορφές, αν έπρεπε να περιμένουμε να συμφωνήσουν όλες οι χώρες, δεν θα είχαμε φτάσει ούτε καν σε αυτά τα δύο μεγάλα δημιουργήματα της Ευρώπης, δηλαδή τη ζώνη Schengen, ξέρετε, ελεύθερη κυκλοφορία, χωρίς ελέγχους, ούτε το ενιαίο νόμισμα. Και για την ενέργεια, ο κύριος Τελόρ έχει την ίδια άποψη. Ε, προσπάθησα κύριε Πρόεδρε να είμαι σύντομος. Μπορούμε, θα μπορούσα να συνεχίσω, θα μπορούσα, αλλά σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ και για μια ακόμη φορά χίλια συγγνώμη που σας ξέχασα. Πέντε λεπτά για τη συζήτηση. Μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις ε, πάνω στο θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Πολύ ενδιαφέροντα όλα σα ακούσαμε. Κάνατε μια ανάλυση νομική για τον κίνδυνο, για την διακυβερνητικό έλεγχο από το Συμβούλιο. Ε, δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος γιατί κάτι λείπει εδώ στην ανάλυση σας αυτό που διδάσκουν οι πολιτικές επιστήμες σήμερα, αυτός που έχει το προσωπικό και, το, και τα χρήματα, τα κονδύλια, είναι αυτός που έχει και την εξουσία. Το 66% όλων αυτών βρίσκεται στα χέρια της Κομισιόν. Ο κύριος Ρομπόη το είπε σε μια, σε μια συνέντευξη ότι δεν έχει την καλύτερη δουλειά. Είδαμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και στο τέλος με την κρίση. Οι, αξιοδο... αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι μεγαλύτερες από αυτές της ε, Κομισιόν. Και τελευταίος, στη δική μου τη χώρα, πολύ περισσότερα νέα είχαμε για την ε, Ισπανική Προεδρία παρά για την Προεδρία του Συμβουλίου. Εγώ είμαι νομικός. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να δίνετε προσοχή στο ποιος έχει την εξουσία και την εξουσία την έχει αυτός που έχει τα χρήματα και το προσωπικό. Ζήτω συγγνώμη για το σχόλιο μου, αλλά δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος για αυτό που λέτε. Ήμουνα δέκα χρόνια εγώ ευρωβουλευτής, γνωρίζω πώς δουλεύουν τα πράγματα και δεν είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει πρόβλημα. Είμαι και μέλος της Ένωσης των Παλαιών Μελών του Κοινοβουλίου αν και τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που, διαβάζουμε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Άλλα ερωτήματα υπάρχουν. Παρακαλώ. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Μονάρ για το νομικό καθεστώς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ποιες πράξεις του Συμβουλίου θα υπόκεινται σε μελέτη του δικαστηρίου αυτό επί της αρχής περιορίζεται σε διαδικαστικές πράξεις. Αλλά όπως είπατε, η διαφάνεια θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για την υποβολή και άλλων πράξεων του Συμβουλίου στο ΔΕΚ και κατά συνέπεια και κάποιων ε, συνταγματικών αρχών όπως ας πούμε θεμελιώδη δικαιώματα ή αναλογικότητα. Ως προς αυτό ποια είναι η απόψή σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το νέο καθεστώς του Συμβουλίου. Είναι ένα αυτόνομο θεσμικό όργανο. Οι, οι αρμοδιότητες του εμπίπτουν στην ε, δικαιοδοσία του α, ε, δικαστηρίου. Βεβαίως ε, υπάρχουν αρκετές προκλήσεις ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για παράδειγμα, αν ε, κάποια προγραμματικά έντυπα όπως αυτό για την ε, περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας θα μπορούσε να είναι αντίθετο με την αρχή της ε, επικουρικότητας. Δεν, αμφιβα... δεν αμφιβάλλω ότι αυτό θα τεθεί ενώπιν του δικαστηρίου για συζήτηση. Θα ήθελα να απαντήσω αλλά να δώσω περισσότερο την απάντηση του δημοσιογράφου για τον, την αξία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ουσιαστικά λοιπόν, πέρα από τις νομικές δυσκολίες, η... αυτό που διαπιστώνουμε από δημοσιογραφικής πλευράς ε, είναι ότι οι αλλαγές είναι ουσιαστικές ε, στις 25 Μαρτίου έγινε μια δήλωση που έγινε η πρώτη συμφωνία για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Ήταν κείμενα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επιπλέον ε, θα μπορούσε να πει κανείς και άλλα πράγματα για τα οποία δεν έχω απάντηση αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, χωρίς να τους αποκαλεί έτσι ήδη συγκάλεσε σύνοδο των ε, αρχηγών ε, κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της, ζώνης, της Ευρωζώνης. Εδώ υπάρχει ε, θέμα προς συζήτηση. πήραν σημαντικές αποφάσεις και μετά όλο αυτό ο μηχανισμός στήριξη για τις χώρες που βρίσκονται σε δυσκολία. Όλα αυτά αποφασίστηκαν όμως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για μας αυτή η νομική πτυχή είναι σίγουρα σημαντική, αλλά είναι δευτερεύουσα σημασία κατά κάποιο τρόπο μπροστά στην πραγματικότητα, διότι οι θεμελιώδεις αποφάσεις λαμβάνονται από μία αρχή η οποία δεν υπάρχει. Ε, το λέγαμε στην ε, στη δημοσιογραφική γλώσσα σύνοδος κορυφής της Ευρωζώνης γιατί δεν υπάρχει σαν νομική έννοια. Βλέπετε λοιπόν ότι όποια και αν είναι η νομική ε, σημασία ενός κειμένου οι αποφάσεις λαμβάνονται όπως πρέπει να λαμβάνονται και να προσθέσει η κυρία Ρώση το ε, 10 έχει πλήρη αρμοδιότητα για τις πράξεις του Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ε, έχουν ε, επίπτωση στους ιδιώτες, αλλά ακόμη και στις περιπτώσεις όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ψηφίζει με πλειοψηφία, μπορεί να υπάρχει ένα κράτος μειοψηφία το οποίο προσφεύγει στο ΔΕΚ για να ζητήσει ακύρωση. Και πρέπει να θυμίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αυτό υπόκειται στην χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή διαφάνεια και όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της εξωτερικής πολιτικής και κοινή ασφάλειας, στην περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί να παρέμβει το ΔΕΚ. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες απαντήσεις, θέλετε να απαντήσετε εσείς. Σε σχέση με αυτό που είπε ο πρώτος ομιλητής, για το, αυτός που έχει τη χρήματα και το προσωπικό έχει την εξουσία που είναι και η Κομισιόν. Εντάξει, σε ένα βαθμό είναι σωστό αυτό που λέει. Αλλά ένα πράγμα που ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι εξαρτάται από ποια οπτική το βλέπει κανείς. Οι περισσότεροι από εσά τους ακαδημαϊκούς θα ξέρετε αυτό που είπε ο Ντόναλτ Πιουκάλα, ότι αν προσπαθήσει κανείς να περιγράψει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν να είναι κανείς σε μια γραμμή, άντρες σε μια γραμμή που προσπαθούν να περιγράψουν έναν ελέφαντα. Κάποιο έπιασε την προβοσκίδα του ελέφαντα και είπε ότι είναι σαφίδι, κάποιο έπιασε το πόδι του και είπε ότι είναι σαν κορμό δέντρου. Κανένα δεν μπόρεσε να δει συνολικά τον ελέφαντα. Οπότε, αν επικεντρωθούμε σε διαφορετικέ πτυχέ τη Ένωση, προφανώ θα δημιουργηθούν και διαφορετικέ εντυπώσει. Αν, α πούμε, δούμε την πολιτική ανταγωνισμού, υπάρχει ισχυρό εκτελεστικό όργανο στον τομέα αυτό. Αν τώρα πάμε στο περιβάλλον, στην περιβαλλοντική νομοθεσία, θα δείτε νομοθεσία από δύο ε, όργανα όπως ε, έχουν οι αρμοδιότητες. Αν πάμε στην εξωτερική πολιτική, πάμε στο Συμβούλιο περισσότερο του οποίου προεδρεύει ο ύπατος εκπρόσωπος. Αλλά εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπει κανείς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς το παρόν ασχολείται με τους τομείς πολιτικής που έχουν να κάνουν με την σύγκληση των εθνικών αρμοδιοτήτων και μέσω ε, ευρωπαϊκών ε, εργαλείων βεβαίω, μέσων και πώ μπορούμε επίση να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση. Οπότε είναι διαφορετικέ απόψει ανάλογα με το πώ το βλέπει κανεί. Το βασικό ερώτημα είναι όλε αυτέ οι αλλαγέ πώ μπορούν να βοηθήσουν. Και αυτό που δεν έχουμε δει είναι πώ βοηθάει η ε, διεύρυνση όλη αυτή την κατάσταση. Η ισορροπία μεταξύ τη διακυβερνητική πλευρά και των υπερεθνικών θεσμικών οργάνων, όπω είπε ο καθηγητή Ρώση, είναι, η κυρία Ρώση, συγγνώμη, είναι κάτι πολύ σημαντικό και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων γύρω από το τραπέζι χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο σήμερα από ό,τι χρειαζόταν πριν από 20 χρόνια για να συζητήσει ένα θέμα. Οπότε κάθε, ε, ένα, κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου μπορεί να ασχοληθεί αποτελεσματικά με το πολύ με δύο θέματα. Παλιά είχαμε πέντε σε κάθε, σε κάθε συμβούλιο. Οπότε, ενώ το ενισχύσαμε έχοντα αυτόν τον ε, πρόεδρο που μπορεί να συντονίσει καλύτερα τι συζητήσει και υπάρχουν και περισσότερε ε, περισσότερα συμβούλια, πιο πιθανό είναι να παραμείνουν τα πράγματα στάσιμα. Ενώ η Κομισιόν μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ καλύτερα τις ε, συνέπειες της, της, της διεύρυνσης. Είναι εδώ μόνιμα, έχουν την θητεία τους, μπορούν για, για πιο μεγάλο χρονικό διάστημα να συζητούν τα θέματα χωρίς να έχουν άλλα προσκόμματα, οπότε αυτό έχει να κάνει με την, με την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ των οργάνων. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να κάνουμε μεγαλύτερη συζήτηση. Είχαμε όμως πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρουσίες ε, από τους έξοχους ε, προσκεκλημένους μας. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη αυτής της τράπεζας για τη συμμετοχή τους και θέλω να σας ευχαριστήσω και σας για την προσοχή σας.